Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κήρυξω την έναρξη της συνεδρίασης. Έχετε σχόλια ή αντιρρήσεις για την και διάταξη. Δεν βλέπω. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι... Α, κύριε Πρόεδρε, την επόμενη εβδομάδα είχε γίνει μια συζήτηση για την ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν θέλω να προτείνω άλλο σημείο στην ημερήσια διάρκεια, αλλά με κάθε σεβασμό θα ήθελα να έχω κάποιες εξηγήσει σε σχέση με τη δήλωσή σας για τα δακτυλικά αποτυπώματα των Ρουμάνων και Βουλγάρων. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συνάδει με το γεγονός ότι είσαστε ένας πραγματικός Ευρωπαϊστής και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τα ίδια δικαιώματα. Χωρίς λοιπόν να χάσουμε πολύ χρόνο, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τι εννοούσατε, γιατί και άλλοι συνάδελφοι μπορεί να θέλουν να το κατανοήσουν. Αυτή η δήλωση πριν από τις διακοπές προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα αγανάκτησης στην Βουλγαρία. Αγαπητέ συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος Μπροκ. Εγώ προσπάθησα και στη Βουλγαρία να το κάνω αυτό σαφές στην επίσκεψή μου. και επίση του συναδέλφου, οι οποίοι με συνάντησαν και θέλησαν να με ρωτήσουν τι ακριβώ έγινε. Αν θέλετε να ξέρετε ποια είναι η θέση μου, μπορείτε να διαβάσετε την ομιλία που έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα καταλάβετε ότι εγώ ήμουνα αυτός ο οποίος ε, εισήγαγε μαζί με άλλους το, πλή, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρξε μία συνέντευξη όπου εγώ επετέθηνα δύο του κυρίου Κάμερον λόγω της ε, δράσης της, Αμερι... της αγγλικής κυβέρνησης που θεώρησα ότι ήταν απόλυτα λανθασμένη και δεν συνείδε με τις συνθήκες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ με 34 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ πάντα έχω υποστηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τόνισα ότι αν θέλουμε να υποστηρίξουμε με αξιοπιστία αυτή την ελευθερία, θα πρέπει τις πολύ περιορισμένες παραβιάσεις που γίνονται να τις εμποδίσουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, αυτό αφορά όλους, ακόμα και τους Γερμανούς. Αυτό το έκανα σαφές. Και πιστεύω ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν κάποιος πηγαίνει σε ένα κράτος και προσπαθεί με καταχρηστικό τρόπο να διεκδικήσει κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνικές παροχές θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό δεν θα γίνει δεκτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Ότι τα άτομα αυτά τα οποία έχουν κάνει πολλαπλές προσπάθειες κατάχρησης των κοινωνικών δικαιωμάτων, ότι έναντι αυτών των ατόμων θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε στα χέρια μας, ώστε να αποτραπεί αυτό στο μέλλον. Και δεν πρόκειται για τίποτα άλλο παρά για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην ε, Γερμανία και την ε, χρήση από τις τοπικές αρχές της Γερμανίας και άλλων χωρών των δυνατοτήτων που τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω λοιπόν να αλλάξω τίποτα σε αυτά που είπα, Σα τόνισα και πάλι ότι υποστηρίζω απόλυτα την ελεύθερη κυκλοφορία, αλλά υπάρχει και το άρθρο της οδηγίας για την οδηγία ε, ελεύθερης κυκλοφορίας το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι ένα άρθρο το οποίο ισχύει ήδη από το 2004 και εξηγεί εκπεφρασμένα ότι όταν πηγαίνει κανείς σε μια άλλη χώρα πότε μπορεί να διεκδικήσει κοινωνικές παροχές και πότε όχι. Αυτό το άρθρο λοιπόν 7 θα πρέπει να εφαρμοστεί για να μην υπάρχουν καταχρηστικές ενέργειες επί τη βάση της ελευθερίας κυκλοφορίας η αγγλική βέβαια στάση είναι απόλυτα απορριπταία γιατί κάνει διάκριση μεταξύ πολιτών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει όμως όλα αυτά τα οποία είπα να δώσουν λαβή σε λαθασμένες ερμηνείες και εγώ χαίρομαι που ο Ρουμάνος ε, Πρωθυπουργός αφού έλαβε τις απαραίτητες διευκρινήσεις έχει ε, θεωρήσει τον εαυτό του ικανοποιημένο σε σχέση με τη δήλωσή μου. Έχετε άλλες παρατηρήσεις. Το κατανοώ κύριε Πρόεδρε. Αλλά υπάρχουν αυτά τα οποία έχουν δημοσιευτεί στις γερμανικές εφημερίδες για τα δακτυλικά αποτυπώματα που πρέπει να γίνονται, να λαμβάνονται για να μην γίνεται η κατάχρηση των κοινωνικών συστημάτων παροχών στις Γερμανίες. Αυτό φαίνει σε σχέση αυτά που είπατε με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά νομίζω ότι αυτά που είπατε είναι εύστοχα και ελπίζω ότι απλώς ήταν μια λαθασμένη είδηση η οποία δημοσιεύτηκε από τις γερμανικές εφημερίδες. Αν διαβάσετε το σύνολο της ε, συνέντευξης στην εφημερίδα Bild, και ίσως μπορώ να σας το δώσω το πλήρως κείμενα, υπάρχει μια αποσπασματική και εσφαλμένη παράθεση αυτών που είπα. Δεν ήταν αυτό το οποίο είπα εγώ προς την κατεύθυνση αυτή, ήταν ακριβώς μια διατύπωση υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας. Γι' αυτό προσκαλώ όλους τους συναδέλφους που τους ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό να έρχονται σε επαφή με τον Πρόεδρο εφόσον το επιθυμούν και τότε μπορεί ο Πρόεδρος να ανασκευάσει αυτά τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Εάν όχι, μπορείτε σε αυτή την περίπτωση να με επικρίνετε δικαιολογημένα. Ακόμα και ο κύριος μιτικόφερ μπορεί να το πράξει αυτό. Έρχομαι τώρα ένα ανακοινώσεις του Προέδρου. Έκανα μια δήλωση τύπου την πέμπτη σε σχέση με την Ουκρανία και ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει υπογράψει ε, διατάγματα και νόμους που κατά την άποψή μας δεν έχουν ε, νομιμότητα. Ήταν 200.000 άτομα στο Μαϊντάν, στην πλατεία δικαιωτική, στο Κίεβο χθε για να διαμαρτυρηθούν. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε μια επικοδομητική εκμετώπιση και σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου σας έχει, ο πρόεδρος μάλλον έχει προσκληθεί σε ένα της Ουκρανίας σε ένα συμπόσιο μαζί με την αντιπολίτευση. Ελπίζω να μην επαναληφθούν οι αντιπαραθέσεις του παρελθόντος. Και φυσικά το γεγονός ότι ο υπέγραψε ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς αυτές τους νόμους δεν εξαίρει ιδιαίτερα την αξιοπιστία του. Και σίγουρα δεν έχει ξεκινήσει αυτή η προβλεπόμενη επίσκεψή μας στην Ουκρανία με καλούς Ιούνους. Όταν έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Βενζέλον, θα επανέλθουμε και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σε σχέση με την Ουκρανία και θα έχουμε την ευκαιρία και πάλι να δούμε ποια ήταν και η εξέλιξη μετά από αυτά τα οποία ζητήσαμε να κάνουν οι Ουκρανικές ε, ε, αρχές. Τρίτη ανακοίνωση για τα, τρίτο σημείο μάλλον για τα πρακτικά. Έχετε κάποιες ε, αντιρρήσεις ή σχόλια για τα πρακτικά. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Εγκρίνονται τα πρακτικά. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα την έκθεση της Doris Park και την έκθεση Προέδρου 2013 για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. μπορώ να σας πω, θα ήθελα μάλλον να μπορούσα να σας πω ότι οι Βόσνοι πολιτικοί είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με γιγάντια βήματα προς την Ευρώπη και είναι ενωμένοι. Δυστυχώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι ένα θέμα για το οποίο και πέρσι και πρόπερσι έχουμε συζητήσει και δεν έχουν επέλθει ιδιαίτερες ε, πρόοδοι. Προσπάθησα φέτος να έχω μια έκθεση πλήρη για τα θέματα αυτά με την ελπίδα ότι θα μπορούσα να καταδείξω ότι υπήρχαν πρόοδοι στη Βοσνία Ζεγοβίνη σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, σε ό,τι αφορά την ε, δικαστική απόφαση του Σάντι Φίντσι και με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιζόταν ίση μεταχείριση όλων των πολιτών στην ε, Βοσνία Ζεχοβίνη και όχι ορισμένα θεωρούνται πολίτες και άλλα θεωρούνται Σέρβοι, Κροάτες κτλ. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δαπανίσει μόνο περιορισμένο χρόνο και προσπάθεια για να πείσει τους ε, ηγέτες της Βοσνίας. 16 ώρες, προηγουμένως 30 ώρες. Μία προσπάθεια λοιπόν να υπάρξει μία διέξοδος από αυτή την κατάσταση αδιεξόδου που υπάρχει στη Σοβία, στη Βοσνία Ζεχοβίνη, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε επίπεδο εκλογικού δικαίου. Εάν δεν γίνει αυτή η τροποποίηση βέβαια, θα είναι προβληματικές και οι επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε λοιπόν τα αποτελέσματα των επικειμένων εκλογών. Έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση επομένως ενώπιόν μας και δυστυχώς η χώρα αυτή έχει πάρα πολλά προβλήματα και όλα περιστρέφονται γύρω από αυτήν την περίπτωση Φίντσι η οποία ακόμα δεν έχει ουσιαστικά επιληθεί. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνουν όλες αυτές τις προσπάθειες που θα κάνουν τη χώρα να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που θέλουν η Βοσνία Ζεγοβίνη να, στην, να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να έχει μια τέτοια αντιμετώπιση σε πολιτικό επίπεδο ώστε να μπορέσει να συνάδει η πολιτική της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών στη Βοσνία Ζεγοβίνη δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται τώρα να τα απαριθμίσω όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να βελτιωθούν τα πράγματα εν γέννη σε σχέση με την εγκληματικότητα. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν συγκεκριμένε δράσει κατά τη διαφθορά στην ε, Βοσνία Ζεχοβίνη σε όλου του τομεί. Στην ε, πολιτική, στι επιχειρήσει, στα μέσα ενημέρωση. Υπάρχει μια ανίερη συμμαχία μεταξύ όλων αυτών σε επίπεδο διαφθοράς. Και πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλε τι προσπάθειε για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικοί θα κατανοήσουν την ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση διαφθοράς. Επίση έχουμε την πίεση που ασκείται εναντίον των αντιπολιτευομένων, αυτών οι οποίοι δεν ακούν την άποψη τη κυβέρνηση. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητε προσπάθειε και σε κρατικό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Και λυπάμαι ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση και τη νεότητα δεν ενεκρίθη για την Βοσνία Ζεγοβίνη, γιατί η χώρα αυτή δεν ήταν σε θέση να δημιουργήσει ένα εθνικό φορέα, ο οποίο θα ήταν ο συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εκπαίδευση και κατάρτισης. Έχουμε το νέο πρόγραμμα Erasmus. Συν θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο προ το συμφέρον των νέων τη Βοσνίας Ζεγοβίνη να μπορούσαν να αντλήσουν κονδύλια οι νέοι από αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει και το θέμα των επενδύσεων στην ε, Βοσνία Ζεγοβίνη. Δεν λειτουργεί κανονικά η δικαιοσύνη, αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει καν σε αυτό το τόσο μικρό κράτος και ένας ενιαίος οικονομικός χώρος. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη βοήθεια ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση για τις οικονομικές μας σχέσεις οικονομικές σχέσεις της Βοσνίας. Έχουν επιληθεί πολλά προβλήματα μεταξύ Κροατίας και Βοσνίας Ερσεγοβίλης. Παραμένει πολλή δρόμος να διατρέξουμε. Υπάρχει και η επιρροή της Σερβίας προς την Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Θα ήταν χρήσιμο να εξηγήσει η Σερβία προς την Ρεπούμπλικα Σέρψκα ότι δεν είναι απόλυτα αυτόνομη, αλλά τμήμα ενός συνόλου που είναι η Βοσνία Ζεχοβίνη. Κάτι άλλο. Ποτέ εγώ δεν ζήτησα από αυτά που έχω διατυπώσει να καταργηθούν φορεί Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο από τις αρχές της Είπα απλώ ότι το γεγονός ότι μετά από τη συμφωνία του Ντέιτον τον η χώρα αυτή είναι διαιρεμένη σε δύο τμήματα, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχτούμε, με την προϋπόθεση ότι τα δύο αυτά τμήματα δεν θα λειτουργούν σαν κρατικές ενότητες, αλλά σαν συνιστώσεις ενός συνόλου, όπως γίνεται με τα ομοσπονδιακά κρατήρια κρατήρια στη Γερμανία. Εμείς θα πρέπει να εμποδίσουμε όμως σε εθνικό επίπεδο να υπάρχει μεμονωμένη δράση. Θα πρέπει να έχουμε κοινού θεσμού, κοινή δικαιοσύνη ένα ενιαίο ανώτατο δικαστήριο. Εγώ φυσικά ποτέ δεν είπα ότι θέλω να υπάρξει διάλυση των συνιστών των κρατών. Και για την Ομοσπονδία στη Βοσνία Ζεγοβίνη έχω πει στην τελευταία συζήτησή μας ότι η μορφή με την οποία έχει δημιουργηθεί αυτή η Ομοσπονδία δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία. Αυτό ήταν ένα σχήμα που προκρίθηκε στην Ουάσιγκτον το 1996 και περιλαμβάνεται στη Συμφωνία της Dayton. Σε δέκα καντόνια είναι χωρισμένη η χώρα. Επιπλέον υπάρχουν δήμοι, επιπλέον υπάρχουν ομοσπονδιακές κυβερνήσεις και επιπλέον υπάρχει και η βοσνιακή αζεγοβινική κυβέρνηση. Όλο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δέκα πρωθυπουργού έχουμε σε αυτό το μικρό κράτο, σε αυτή τη μικρή ομοσπονδία. Σε κάθε... Έχουμε δέκα υπουργού ε, παιδείας και κατάρτισης σύν τον ομοσπονδιακό υπουργό. Πώς περιμένετε ότι θα λειτουργήσει ένα τέτοιο κράτος. Γι' αυτό λέμε ότι όλη η διοίκηση στη Βοσνία Ερσεγοβίνη θα πρέπει να ορθολογικοποιηθεί, θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα και θα πρέπει να είναι πολύ λιγότεροι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να λειτουργήσει ένα τέτοιο σχήμα όταν το ένα επίπεδο παρεμποδίζει το ανώτερο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα οποία έχουμε ε, δει στην χώρα αυτή τη Βοσνία Ζεγοβίνη. έχω επίσης ε, περιλάβει πολλές συστάσεις συναδέλφων οι οποίοι θέλησαν να καταθέσουν τροπολογίες στην έκθεσή μου. Κάναμε μια κοινή εργασία για να καταλήξουμε σε 16 τροπολογίες συμβιβασμού. Και έχουμε κρατήσει το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο στο πρίο, κοντά στο Πρίοντορ ανακαλύφθηκε ένας μαζικός τάφος στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα. Το έχουμε συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο στην έκθεση, γιατί αυτό ανήκει στην ιστορία και στην αποκατάσταση της αλήθειας. Επίσης στην περίπτωση Νταμιάνοβιτς, που ήλθε ενώπιον του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτό είναι σημαντικό για τις μελλοντικέ ε, αποφάσεις που θα ληφθούν σε περίπτωση τέτοιου είδους αδικημάτων. Παραμένει το γεγονός, όπως αναφέρεται στην έκθεση, ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγνοωμένων επίσης. Υπάρχουν πολλά προβλήματα για την επιστροφή των ε, προσφύγων. Δεν μπορούν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν να το πράξουν. Έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά είναι πάρα πολλά τα οποία παραμένουν να γίνουν. Και τόνισα ότι η Βοσνία Ερσεγοβίνη έχει περιοχές οι οποίες όπως η Κοσοβίνα που είναι ερημωμένη όπως αμέσως μετά τον πόλεμο της ε, Βοσνίας του 1996 όπου δεν μπορεί κανείς να γυρίσει, όπου οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν σε κανένα να επιστρέψει, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ξαναχτίσει κανείς τα σπίτια του και να έχει πρόσβαση σε ρεύμα, νερό κτλ. Λείπει η καλυφέληση από πάρα πολλούς, σε πάρα πολλούς χώρους και αυτό νομίζω το τονίζει η έκθεσή μου. Δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει διαφωνία των συναδέλφων με αυτή την έκθεση, το βασικό στοιχείο της. Έχουν προσθέσει πολλά συνάδελφοι, έχουν τονίσει ορισμένα σημεία, δεν θέλησαν να απαλύνουν πολλά αυτά, τα οποία λέω. Και τα βασικά προβλήματα είναι καταρχήν το πρόβλημα της ε, συνταγματικής αλλαγής, το θέμα της ε, διαφθοράς, το θέμα της λειτουργίας της δικαιοσύνης, ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης, η κατάρτιση και η δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου. Η περιφερειακή συνεργασία, όπως σας είπα, είναι καλή. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα δεν έχει επιληθεί για την Βοσνία Ζεχοβίνη. Είναι η μόνη χώρα που δεν επιτρέπει την είσοδο Κωσοβάρων σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν το καταλαβαίνει αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Κόσοβο και ανήκουν στη βοσνιακή μειονότητα δεν μπορούν να πάνε στην πατρίδα τους γιατί η βοσνιακή κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι να πάνε στη Σερβία, μεν, αλλά όχι στη Βοσνία. Αυτό δεν βγάζει κανένα νόημα. Και εν κατακλείδη θα ήθελα να πω κάτι το οποίο το λέω με μεγάλη σοβαρότητα. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση είχα κάνει μια έκκληση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο αρχικό κείμενο και στους Υπουργούς Εξωτερικών. Να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία τους στη Βοσνία Ζεγοβίνη, να καταδεικνύουν περισσότερο ενδιαφέρον για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Δεν αρκεί να είναι εκεί παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και όταν πηγαίνει η Λέδη Άστον, πηγαίνει εκεί η, η Παλίτς, Παρά το γεγονός ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αλλά το να πηγαίνει ένας Πρωθυπουργό και να. Αν μπορεί να πηγαίνει ένα Πρωθυπουργό και να μιλάει στη Βοσνία Ζεγοβίνη και να μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω έχει γίνει στην περίπτωση τη Σερβία, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να τα κάνει όλα η Κομισιόν και θα μπορέσει και ο λαό τη Βοσνία Ζεγοβίνη να πιστέψει ότι δεν του έχουμε λησμονήσει τελείω. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει και μια πολιτική παρουσία και όχι μονάχα η Κομισιόν. Θα πρέπει να δείξουμε το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Βοσνία και να τους πούμε ότι φτάνει, πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες μεταλλαγές και τροποποιήσεις και στη χώρα τους. Αυτά λοιπόν θέλω να πω εγώ. Ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τις συμβαστικές τροπολογίες και θα έχουμε μια καλή ψηφοφορία αύριο για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Επτά ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο και έχουμε κάποιες εκθέσεις ακόμα να εξετάσουμε. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω κάποια... Εννέα είναι τώρα συνάδελφοι που θέλουν να λάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ να αυτοπεριοριστείτε και να ερωτήσετε τον εαυτό σας αν αξίζει τον κόπο να λάβετε το λόγο γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στους επόμενους ομιλητές. Έχουμε λοιπόν 1,5 λεπτό. Είμαι γενναιόδο. 1,5 λεπτό λοιπόν για τον κάθε ομιλητή, Άννα Γκόμης. Θα μιλήσω εκ μέρου τη ε, Μινέα Μποκούτ, τη γιατριά μα, η οποία δεν μπορεί να είναι εδώ τώρα και ζητά συγγνώμη. Σε ό,τι αφορά την έκθεση πρόοδου, βλέπουμε ότι δεν ήταν τεράστια η πρόοδο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη το 2013. Δεν είναι καινούριο να λέμε ότι καθυστερεί σε σχέση με του γείτονε και την όλη περιοχή η χώρα αυτή στην διαδικασία προσχώρηση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ομάδα πιστεύει ότι η διαδικασία προσχώρηση τη Βοσνία Αρζεγοβίνη θα πρέπει να γίνει μια προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι καθοριστικό στοιχείο για την ειρήνη και τη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων. Υπό αυτήν την οπτική γωνία δεν κατανοούμε και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω την εισηγητριά μα, την κυρία Πακ, γιατί τοποθετείται αρνητικά ως προς την τροπολογία 6 την δική μας. Εκεί όπου τονίζεται ότι η προοπτική της ευρωπαϊκής προσχώρησης θα πρέπει να προσφερθεί στο σύνολο της χώρας, σε μια ενιαία δηλαδή Βοσνία Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Μόνο έτσι μπορούμε να το αντιληφθούμε. Επίσης πιστεύουμε ότι το να συνεχιστεί αμύωτη δέσμευση από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και περισσότερη ε, δέσμευση από τους ε, αρχηγούς κατών και κυβερνήσεων και υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν καλοδεχούμενο. Για τις μεταρρυθμίσεις πιστεύουμε ότι οι εκλογές του 2014 ούτως ή άλλως πλησιάζουν γοργά και θα πρέπει η Βοσνία Ζεγοβίνη να επιταχύνει την υλοποίηση της απόφασης ΦΙΝΤΣΙ επιφερόντας τις ανάλογες, ε, τις απαιτούμενες αλλαγές των εκλογικών νόμων προκειμένου να διεξαχθούν αυτές ομαλά. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε αναγκαίο να μετατραπεί η Βοσνία Ζεγοβίνη σε ένα αποτελεσματικό και πλήρως λειτουργών κράτο. Αυτό θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα για τους πολιτικούς ε, ηθήνοντες τη χώρα. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, θα πρέπει να είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες της Βοσνίας Ερσεγοβίνης κατά την ομάδα μας και γι' αυτό καλωσορίζουμε την ε, ε, στήριξη των υπόλοιπων ομάδων στην τροπολογία 72, τη δική μας τρία, προκειμένου να στηριχθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Βοσνία Ζεγοβίνη και να υπάρξει και τεχνική αρρωγή σε αυτό το θέμα με την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας εκεί. Ε, εν είδη συμπεράσματο, νομίζουμε ότι συντάχθηκε μια έκθεση που δείχνει ότι υπάρχει δέσμευση μεν προ την διαδικασία προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ποσνία Ριζεγοβίνη, αλλά από τη χώρα αυτή και του ηγέτε τη περιμένουμε να μα φέρουν και πιο απτά αποτελέσματα. Και όχι για το δικό μα όφελο, αλλά για την ευημερία των πολιτών τη χώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κορνέλισεν είναι σωστή προφορά. Ευχαριστούμε την κυρία Πακ για μια ισόρροπη έκθεση που είναι κάπως λιβερή αλλά έτσι είναι και η κατάσταση. Με μεγάλη μου θλίψη έχασα την ε, συνάντηση για την εξέπρεση συμβαστικών λύσεων, δυστυχώς, αλλά ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που συμπερίλαβαν κάποιες από τις προτάσεις μου. Θα συμφωνήσω με όλες τις παρατηρήσεις που έκανε η κυρία Πακ μόλις τώρα η έλλειψη πρόοδου της Βοσνίας Ζεγοβίνης είναι πραγματικά πολύ ε, θλιβερή. Θα πρέπει οι πολιτικοί ε, να ξαναεξετάσουν ε, τα δικά τους συμφέροντα και τον, τις μελλοντικές προοπτικές της δικές τους και των πολιτών της χώρας. Νομίζουμε ότι οι συμβαστικές λύσεις είναι πολύ εύστοχες, ιδίως η τρίτη, που ζητά από να επιταχύνει τις προσπαθίες της και να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα. Κάποιες φορές φαίνεται ότι Υπάρχουν κατεπήγοντα τι προτεραιότητε τη διεθνού κοινότητα άλλου είδου και η Βοσνία Ζεγοβίνη ουδέποτε αποτελεί μια από τι πρώτε προτεραιότητε. Για τη συμβαστική λύση 11 τώρα. Εκεί λέγεται και να εγγυηθούμε ίσα δικαιώματα για όλου του ε, συμμετέχοντες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, της σερβικής Αυτό όμως δεν ε, συνάδει με το πνεύμα της απόφασης SDT. Finch. Θα πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν εδώ, τι γίνεται με τα ριδιοτηλόραση και τα δημόσια μέσα επικοινωνίας. Τελευταία παρατήρηση για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι βεβαίως μείζον ζήτημα, κάτι που θα πρέπει να το χειριστούμε ως προτεραιότητα. Μεν, και στην προφορική τροπολογία παρόλα αυτά λέγεται ότι θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι κάτι είναι απόλυτη προτεραιότητα. Absolute priority. Ίσως αν διαγράφαμε τον όρο absolute, απόλυτη προτεραιότητα, να ήμασταν περισσότερο σύμφωνοι με όλα αυτά. Παρακαλώ. Δώστε καλό παράδειγμα κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ. Μια ισορροπημένη, συμπαγής έκθεση που αναφέρεται στην κατάσταση στη χώρα με ικανοποιεί ο θετικό τόνο τη έκθεση. Ο εκλογικό νόμο είναι σημαντικό, όπω είπε και η κυρία Γκόμε. Οκτώβριο 2014 θα έρθει και ο εκλογικό νόμο θα πρέπει να είναι έτοιμο. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή δίνει το πιο σημαντικό μήνυμα, ότι δηλαδή είναι η πολιτική ελίτ και όχι ο κόσμος που είναι υπεύθυνη για την κατάσταση. Ο συντονισμός ε, του μηχανισμού είναι κάτι πολύ βασικό. Πρέπει οι διαπραγματεύσεις να γίνονται με μία φωνή από την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να ενισχυθεί. Στη Μπάνια Λούκα, στην ε, Δημοκρατία της Έρσπρα, ακούμε ότι με την έκθεση αυτή θα πιέσουμε τους πολιτικούς προκειμένου να δικείται πιο κεντρικά η χώρα. Δεν είναι αλήθεια. Εγώ διάβασα την έκθεση και αυτό που κάνει η κυρία Πάκη είναι ότι ζητάει συνταγματικέ μεταρρυθμίσεις, προκειμένου όμως η χώρα να λειτουργεί καλύτερα και να έχει λιγότερο διοικητικό άχθος. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα. Καλά ήταν, κύριε Κούκαν. Ο κύριος Στύρ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Βοσνία Αρζεγοβίνη έχει βαλτώσει η κατάσταση. Και γιατί δεν φταίνε ούτε οι Κροάτες, ούτε οι Βόσνοι, ούτε οι Σέρβοι, ούτε φυσικά οι κάτοικοι της Βοσνίας Αρζεγοβίνης. Πού οφείλεται η βάλτωση αυτή. Από τη μια μεριά υπάρχουν οι αποσχιστικές τάσεις και από την άλλη μεριά υπάρχει η κεντρική δίκηση, η ενίσχυση αυτής της κεντρικής δίκησης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η συνάδελφος Ντόρις Πακ στην τροπολογία αριθμός 19 αναφέρει την αναγκαιότητα να τονίσουμε περισσότερο την σημασία που έχει να συνεχίσουμε στον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ομοσπονδιακό δηλαδή επίπεδο. Εγώ υπογραμμίζω στις τροπολογίες ότι ο φεντεραλισμό είναι κάτι πολύ βασικό για την Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και γι' αυτό και εγώ όπω και η συνάδελφος Πακ και μένα μου επιτέθηκαν διάφοροι από την Ρεπούμπλικα Σέρφκα, μάλλον τα μέσα ενημέρωσής τη, μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, κάποια ριζοσπαστικά μέσα ενημέρωσης της Ομοσπονδίας που ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την πρόοδο της χώρας προκειμένου να ενταχθεί αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αυτό είναι το στοιχείο κλειδί. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να εξυπηρετεί τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Νομίζω ότι οι σεβαστικές τροπολογίες τελικά περιλαμβάνουν και αυτό που με ενδιαφέρει μεν ιδιαίτερα, ο φεντραλισμός δηλαδή. Στη συμβαστική 12 δεν πρέπει να μιλάμε για segregation, για τέτοια διάκριση, αλλά να τονίζουμε την πρόοδο που έχει πετύχει η Βοσνία Ερζεγοβίνη και που επιτυχάνεται μέσω της ομοσπονδιακής διάστασης. Οι επιθέσεις εναντίον αυτού δείχνει ότι δεν είναι όριμη η κατάσταση μερικές φορές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πίκολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την συνάδελφο Δόρις Πακ. Το 2013 ήταν ευνοϊκή κατάσταση. Η Κροατία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει χίλια χιλιόμετρα σύνορα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Άρα υπάρχει ευρωπαϊκό σύνορο. Όμως το θέμα πάει πέρα από τα σύνορα. Παρόλο που το γεγονός αυτό αποτελεί κάποιο κίνητρο. Μετά πάντως από διάφορους γύρους διαπραγματεύσεις και μετά από τις διαπραγματεύσεις που έκανε ο Επίτροπος Φίλε για ενδεχόμενη ένταξη, βλέπουμε ακόμα να μην προχωράμε πολύ. Ενώ οι προσδοκίες είναι τεράστιες στη χώρα αυτή. Η χώρα αυτή βρίσκεται σε μια χρόνια βάλτωση Πρέπει λοιπόν να κάνουμε έκκληση στους πολιτικούς στη Βοσνία Ερζεγοβίνη προκειμένου να αρχίσουν να δουλεύουν ειλικρινά προς το όφελος των ίδιων των πολιτών τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριο Βουλιάνικ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την κυρία Πάκ για την ισορροπημένη και αρεαλιστική αλλά και φιλική έκθεσή τη. Και το τονίζω το φιλική γιατί προσπαθεί να βοηθήσει τη χώρα προκειμένου να λειτουργεί κανονικά, φυσιολογικά. Οργανώνεται βάσει το στοιχείο της ειρηνευτικής ε, συμφωνίας που όμως πια δεν φτάνει για να οργανώσει τη χώρα και πρέπει να υπάρξουν ε, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις όπως προτείνει η έκθεση της κυρίας Πακ. Δεν ονειρεύομαι και δεν νομίζω ότι κανένας άλλος έχει ψευδεστήσεις δεν μπορούμε εμεί να πούμε στον κόσμο τη Βοσνία Ερζεγοβίνη τι είδου ομοσπονδία πρέπει να έχουν, τι είδου χώρα πρέπει να φτιάξουν. Αυτό είναι δικιά του δουλειά. Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν μόνοι του, όχι εμεί. Αλλά πρέπει να το αποφασίσουν ότι θα έχουν μία χώρα, ενιαία, Όπω και αν είναι αυτή η χώρα. Υπάρχουν εκατοντάδε προβλήματα με εκατοντάδε διαφορετικέ στάσει από του διάφορου υπουργού και υπάρχει μια πολιτική ελίτ η οποία δεν δέχεται σε βιβασμού δεν θέλει να προχωρήσει σε συμβασμούς για να λειτουργήσει η χώρα. Πρέπει όμως να υπάρχει μια συνένεση όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και στα υπόλοιπα συμβιβασμοί. Υπάρχει ένα τμήμα της έκθεσης με το οποίο δεν συμφωνώ. Λέει η έκθεση ότι οι ιδιωτικοποίησεις πρέπει να επιταχυθούν στη χώρα. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που χρειάζονται. Έχουν αρκετά προβλήματα χωρίς τις ιδιωτικοποίησεις προβλήματα με τη διαφθορά, με το οργανωμένο έγκλημα, με το λαθρεμπόριο. Δεν χρειάζονται κι άλλο ένα πρόβλημα τώρα με μια ευρία ιδιωτικοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κοπά. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Να συγχαρώ την κυρία Πάκ για την εξαιρετική έκθεση που συνέταξε και νομίζω για την, για την υπάρχει ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο. Κάποιε σύντομε παρατηρήσει. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανικανότητα των πολιτικών εθνοτών τη χώρα να καταλήξουν σε μια κοινή θέση. Νομίζω ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε το πρόγραμμα μια ενιαία Βοσνία Ζεγοβίνη, ούτε του πολίτε τη. Και συμφωνώ με τον κύριο Κούκαν σε ό,τι μόλι είπε. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στι συνταγματικέ μεταρρυθμίσει και να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή απευθεία με την κοινωνία των πολιτών. Εάν οι πολιτικοί δεν είναι στο ύψο των περιστάσεων, εάν δεν μπορούν να φτάσουν στο ύψο τη φιλοδοξία μια ενίας και ευρωπαϊκής Βοσνίας. Πιστεύω ότι οι πολίτες της χώρας αυτής τουλάχιστον το επιθυμούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπροκ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την έκθεσή της. έχει προσφέρει τη στήριξή της στη Βοσνία Ζεγοβίνη ε, στην κατεύθυνση της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω, ε, και εγώ αλλά πιστεύω και όλοι οι Κροάτες συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου, ότι δεν πρέπει να υπάρξει ιστορική αδικία με διάκριση κατά της Βοσνίας Ζεγοβίνης. Δεν θέλουμε να γίνει ο τελευταίος τροχός της αμάξης ε, ως προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα αυτή. Η συμφωνία λοιπόν ε, σύνδεσης και συνεργασίας δεν έχει τεθεί σε ισχύ και Νομίζω ότι η απόφαση σας Διτσβίντσι θα πρέπει να ερμηνευτεί ως εξής. Θα πρέπει να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε ισότητα και συνταγματική ε, ίση μεταχείριση των ε, Σέρβων πολιτών, διότι είναι ε, ένας από τους βασικούς πληθυσμούς της χώρας αυτής, αλλά το ίδιο και για τους Κροάτες. Θα πρέπει λοιπόν να πω ότι είναι κρίμα που ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης της Βοσνίας Ζεγοβίνης ανεστάλλει προφανώς υποβαθμίζει και κάπως ε, παρεμποδίζει το, την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Δυσκολεύει την επίτευξη περαιτέρω πρόοδου. Συζητώντας με την πολιτική ηγεσία της Βοσνίας Ζεγοβίνης, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει κατάλληλο συντονισμός για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη χώρα. Ακόμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει στην επίλυση κάποιων από τα εκρεμή ζητήματα, όπως το πρωτόκολλο για τη Συμφωνία ε, Σταθεροποίησης και Συνεργασίας με την Κροατία, αλλά θα θέλαμε και συνομιλίες με την ε, κυβέρνηση στη Βοσνία για να ε, υπάρχουν υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στα δηληστήρια της χώρας που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία πολλών πολιτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια. Αλλά πρέπει να πω ότι και εγώ είμαι απόλυτα απογοητευμένη για τα αρνητικά αποτελέσματα της συνάντησης προηγούμενης Παρασκευής στο Σαράγεβο. Είναι φανερό ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί καμία λύση. Δηλαδή δεν υπήρξε καμία πολιτική θέληση για να γίνει κάτι τέτοιο. Έχω πει ήδη στο παρελθόν στο Σαράγεβο ότι το θέμα της αναγνώρισης των εκλογών θα παραμείνει εκρεμές αν δεν επιληθεί το θέμα της υπόθεσης Σέντιτς Φίντζη. Θα πρέπει να ενδιαφέρεται η δημοκρατία της Βοσνίας Ερσεγοβίνης για όλους τους ε, πολίτες της και κάνω μια έκκληση προς την εισηγήτρια και στην ομάδα μου να είμαστε παρόντες στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Όχι μονάχα παρόντες, αλλά να μπορέσουμε εκεί να έχουμε μια ενιαία φωνή ως Ευρωπαίοι. Θέλω φυσικά να χαιρετήσω το γεγονός ότι η πρόσφατη έκθεση της Frontex δείχνει ότι πέρσι και προηγουμένως, τον προηγούμενο έτος έχει μειωθεί ο αριθμός των ετούντων άσυλο από τη Βοσνία Ζεγοβίνη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πρέπει όλα να, να γίνουν ώστε να μην ε, υπάρξει αναστροφή αυτού του κλίματος στην περιοχή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί εξακολουθούν να δακτυλοδεικτούν τους πολιτικούς. Μα σε μια δημοκρατία όπως η Βοσνία Ζεγοβίνη, ποιοι εκλέγουν τους πολιτικούς ή ο λαός. Ο λαός εκλέγει τους ηγέτες που θέλει. Αν έχουμε δυσκολίες με τους ηγέτες, αυτό είναι και μια απόφαση του ίδιου του λαού. Παρ' όλα αυτά εγώ χαίρομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα την επιμονή και την υπομονή της Doris Park και την αφοσίωσή της για τα θέματα αυτά, εγώ ήμουν κάπως σκεπτικιστή σε σχέση με τη συμφωνία του Dayton, γι' αυτό δεν μπορώ να πω ότι απογοητεύομαι τελείως με την έλλειψη ενότητα στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Θα απογοητεύομαι περισσότερο αν γινόταν κάτι αντίθετο. Μετά από τον εμφύλιο πόλεμο όμως είναι γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χώρα η Βοσνία Ζεγοβίνη και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει να γίνει κάποτε μια ενιαία χώρα είναι ακόμα μία ομοσπονδία και θα είναι πάντα μια ιδιαίτερα αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Ίσως με το παράδειγμα του Βελγίου. Γιατί η ιδέα του να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση στο Σαράγεβο αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει πραγματικότητα λόγω των διαφορετικών απόψεων των συνιστώσεων ομάδων. ομάδων. Αλλά από άποψη Realpolitik η ομάδα μου υποστηρίζει την έκθεση, υποστηρίζει τις τροπολογίες και φυσικά υποστηρίζουμε τη Βοσνία Ζεγοβίνη ως μελλοντική υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό να γίνει μια υποψήφια χώρα, αλλά δεν θέλω αυτή τη στιγμή να, έχω προσδοκίες οι οποίες κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν. Ένα πράγμα για το οποίο συμφωνώ είναι σε σχέση με αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της ΚΟΕ, δεν βλέπω την αντίστοιχη παράγραφο, αλλά αν πράγματι υπάρχει μια έκκληση για περισσότερη απορρίθμιση και ιδιωτικοποίηση, για μένα θα ήταν καλό αυτό. Αλλά δεν βρίσκω την παράγραφο που να τα λέει αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, για μένα η έκθεση ΠΑΚ είναι πάρα πολύ οργανωμένη για την αντιμετώπιση διαφθορά οργανωμένου εγκλήματο, καλύτερη διοίκηση, προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν πια τη χώρα αυτή προ την κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προσδοκιών της. χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει πρόσωπος της Κομισιόν και εμείς συμφωνούμε ιδιαίτερα με την εισηγήτρια σε σχέση με την ανάλυση της πολιτικής κατάστασης, ιδίως την ε, δήλωση αυτή για την ε, ευρωπαϊκή της προοπτική. Υπήρξε περιορισμένη πρόοδος σε ό,τι αφορά τον οδικό χάρτη για την ε, πρόοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξε ιδιαίτερη συζήτηση με τη Βοσνία Ζεγοβίνη για την εφαρμογή της απόφασης Σέντιτς Φίντσι και επίσης για την προσαρμογή μετά από την ε, ένταξη της Κροατίας. Για την εφαρμογή της απόφασης Σέντιτς Φίντσι, όπως ξέρετε, συνεχίζονται οι προσπάθειες. Η Κομισιόν έχει περάσει ακόμα μια νύχτα χωρίς απτά αποτελέσματα, αλλά συνεχίζει να βοηθάει τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Είναι πολύ σημαντικό να επιληθεί αυτό το θέμα γιατί κάνει σαφώς, κάνει σαφή τα κάνει σαφής μάλλον τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τους εταίρους μας στην ε, Βοσνία Ζεγοβίνη και από αυτή την άποψη η τροπολογία επαριθμών 3 η οποία ζητά τη συνεχιζόμενη δέσμευση των ευρωπαϊκών θεσμών και σίγουρα αυτό θα γίνει από την Κομισιόν και των διεθνών φορέων είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη δική μου άποψη. Κάτι ακόμα για την προαντεξιακή <clears throat> χρηματοδότηση, την ΕΠΑ. Η Κομισιόν ενέκρινε πριν από τα Χριστούγεννα ένα πρόγραμμα 42 εκατομμύριων ευρώ εστιασμένο σε ορισμένου τομεί, κάπω λιγότερο από αυτό το οποίο προβλεπόταν, με στόχο να υποστηρίξει τι ανάγκε των πολιτών, του Ρωμά, την ανάγκη δικαιοσύνη κτλ. Αυτό που μα ενδιαφέρει περισσότερο όμω και το οποίο είναι σαφέ στην έκθεση είναι η ΕΠΑ 2 όπου δεν έχουμε ακόμα τη βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε συντονισμό με τους εταίρους μας για να προετοιμάσουμε σε επίπεδο διαλόγου την ΕΠΑ 2. Αυτός ο διαφθορμένος λοιπόν διάλογος που θα έχετε με τον Επίτροπο κύριο Φίλε για την ΕΠΑ θα πρέπει να σας δώσει τη δυνατότητα να δούμε πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την προενταξιακή αρρωγή προς την Βοσνία Ζεγοβίνη. Πάρα πολύ σύντομα, λέει η κυρία Πακ, δεν είναι παρούσα η κυρία Γκόμες, ίσως μπορούν οι συνάδελφοί της να της το πούν αυτό. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για το περιεχόμενο. Απλώς λέει η κυρία Γκόμες και πάλι αυτό το οποίο λέω στην πρώτη μου τροπολογία. Έχω τροποποιήσει το σημείο μου α. Λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προσφυλωμένη στην δυνατότητα προσχώρηση τη Βοσνία Ερεγοβίνη. Το αλλάζω αυτό λέγοντα ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έντονα, στεναρά υποστηρίκτρια μια ε, ενιαίας Βοσνίας Ζαζεγοβίνης και της ε, προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο στεναρό από αυτό που είπε η κυρία Μπόσκουρτ. Η κυρία Μπόσκουρτ με τη δική της τροπολογία έχει κάνει κάποιες ε, αναφορές στην Βοσνία και το Κωσυφοπαίδιο. Αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε κατά μέρο. Θα πρέπει να κρίνουμε τη Βοσνία ως έχει και όχι σε σχέση με θέματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την εσωτερική κατάσταση στη Βοσνία. Δεν είμαι εναντίον λοιπόν του να υπάρχει μία χώρα. Λέω μια ισχυρή, κυρίαρχη και ενωμένη χώρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Είμαι εναντίον της πρωτοπολογίας της κυρίας Γκόμες μόνο αν δεν γίνει δεκτή η δική μου, λέει η κυρία Πάκ. Πάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, και ο κύριος Βροκ. που είναι το θέμα της έκθεσης προόδου για την μου με εισηγητή τον κύριο Χάουιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία Πακ και εγώ είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ποτέ δεν είμαστε σε ανταγωνισμό μεταξύ μας. Πρέπει να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στη χώρα για την οποία είμαι εγώ αρμόδιος. Πρώτον, όπως και πέρυσι, προτείνω οριζόντιες τροπολογίες. Με μία μνήα που γίνεται στον ε, τίτλο της χώρας, «Στέως Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και μέσα αναφέρεται η Μακεδονία, οι Μακεδόνες, κάτι το οποίο ενέκρινε και η Επιτροπή και συνάδει με τα Ηνωμένα Έθνη οτιδήποτε άλλο θα χρησιμοποιώ λέξεις όπως η χώρα κλπ. Και όχι τον τίτλο, ακριβώς για να αποφύγουμε να υπάρχει αντίφαση και να παίξουμε πινκ-πονγκ με το όνομα, κάτι που έγινε πέρυσι. Τώρα, όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες, οι δύο ζητάει από την Ελληνική Προεδρία πολλοί συμφωνούν μαζί μου ότι ζητάμε από την Ελληνική Προεδρία να μας βοηθήσει ο κύριος Κυρίλοφ με βοήθησε στη διατύπωση του κειμένου για το ότι η έναρξη συνομιλιών θα βοηθήσει την πρόοδο ότι μερικές φορές, όπως είπε και ο κύριος Κόβετς, κάποιες ε, πολιτικές δημιουργούν πρόβλημα. Υπάρχει και η Συμβαστική τριά, που αναφέρεται στην τρέχουσα κατάσταση των μεταρρυθμίσεων, της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων. Στη συμβαστική μου δέχτηκα τη διατύπωση του κυρίου Σαλαβράκου, την τροπολογία του δηλαδή, για το ότι πρέπει να τηρηθούν όλα τα κεκτημένα Αλλά συμπληρώνω εδώ και με τη δικιά μου τροπολογία που λέει ότι υπάρχει όμως ένας μεγάλος βαθμός ευθυγράμμισης στα κεκτημένα. Τέσσερα, όσον αφορά τις σχέσεις καλής γυτνίασης. Εγώ να δεχτώ της κυρίας Κοπά την τροπολογία που λέει κατά προτίμηση να λυθεί το θέμα του ονόματο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Εντάξει, ναι, ελπίζω το Κοινοβούλιο να δεχτεί την πρόταση του κυρίου Φίλου ότι θα μπορούσε να εξεταστεί αφού αρχίσουν οι συνομιλίες. Αλλά το κατά προτίμηση που λέει η κυρία Κοπά είναι κάτι που μπορώ να στηρίξω. Για τα αποτελέσματα και λοιπά και της κυρίας Γιαννάκου και του κυρίου Πίκολα τις τροπολογίες για τον όρο essential, ουσιαστικές. Συμβιβαστική 5 τώρα, σε σχέση με το θέμα του ονόματος. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και παλιότερα, δηλαδή να λέμε ότι τα διμερεί ζητήματα δεν παίζουν ρόλο στη διαδικασία ένταξης, αλλά για το θέμα του ονόματος μπορώ να δεχτώ για τον κύριο Κουμτσάκο και Πίκολα που λένε ότι η πρόοδος είναι ζωτικής σημασίας και ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που γίνονται ακόμα και αν είμαστε επικριτικοί στην διαδικασία. Εδώ ακολουθούμε τις προτάσεις Κόπα και Κούκαν αναγνωρίζουμε επίσης την ε, ανάγκη για πραγματική πρόοδο. Όσον αφορά την συμβαστική τροπολογία 6 τώρα, πάλι για το όνομα Δεχοβούλινετς και Κουμτσάκου τροπολογίες, για να επιτευχθεί πρόοδος χωρίς άλλη καθυστέρηση. Να χρησιμοποιήσουμε τον όρο efforts, προσπάθειες. Να αναφερθεί η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, όπως πρότεινα η κυρία Κοπά, και η κυρία Γιαννάκου προτείνει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και η χώρα η και άλλοι πρέπει εκ των προτέρων να εξηγούν τα πλεονεκτήματα από την επίλυση του ζητήματος του ονόματος. Συμβαστική 7 τώρα. Θέλετε να συνεχίσω μία-μία τροπολογία μου να σας εξηγήσω ή Λοιπόν, έρχομαι στη συμβαστική 7 για τα θέματα με τη Βουλγαρία. Εδώ ακολουθώ τις διατυπώσεις Κυρίλοφ, Γιούτσεβε και Ήλτσεφ. Κυρίως προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρα συμφωνία, in due time. Από τα ιστορικά επιχειρήματα, εδώ ακολουθώ τις τροπολογίες Κόρατσοφ και Κίλντοφ και ελπίζω ότι θα θεωρήσουν ότι σωστά αντικατοπτρίζεται το πνεύμα των τροπολογιών του συμβαστική αυτή. Όσον αφορά τώρα την συμβαστική τροπολογία, ναι, για τις εκλογές εδώ, θέλω να κρατήσω κυρίως την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της ΟΑΣΕ για εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Εδώ ακολούθησε διατύπωση του κ. Σαλαβράκου και άλλων. Και αναφέρομαι σε ανεξάρτητη υπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων. Και όσον αφορά τα θέματα τα οποία παραμένουν, εδώ ακολούθησα την διατύπωση Τάνοκ και του κ. Βούριονιτς για τους εθνικισμούς. Εδώ δεν κατηγορείται ούτε χώρο ούτε κανένας στη χώρα για εθνικισμό. Απλώς λέει ότι ο εθνικισμός είναι κάτι με τον οποίο διαφωνούμε γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για οποιαδήποτε χώρα. Ο εθνικισμός καμιά φορά μπερδεύεται με τον πατριωτισμό και ο πατριωτισμός είναι κάτι τελείως διαφορετικό και θετικό. Εξού και αυτή η τροπολογία. Όσον αφορά τις γλώσσες, κάτι άλλο το οποίο δημιουργεί ανησυχίες. Η χώρα δεν θέλει βέβαια να φύγει ο όρος Μασεντόνιαν από την ορολογία. Η τροπολογία αυτή, αυτό που κάνει, είναι ότι αναφέρει την επιθυμία των διαφόρων εθνοτήτων να μάθουν ένα στη γλώσσα των άλλων. Να υπάρχει μια δίγλωση εκπαίδευση, όπως λέει η κυρία Κορνέλισον και η Πράσινη. κοιτάμε το θέμα της αρχής και ενθαρρύνουμε την εκμάθηση της γλώσσας του άλλου. Νομίζω ότι η συμβαστική αυτή τροπολογία είναι δίκαια, θετική και επικοδομητική. Το θέμα των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης, αυτό ίσως είναι το πιο καυτό, το πιο δύσκολο θέμα. Η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης πέρασε στις 26 Δεκεμβρίου και υποβλήθηκαν και τροπολογίες από το Κοινοβούλιο της χώρας την προηγούμενη εβδομάδα και θα εξεταστούν αυτή την εβδομάδα. Οπότε εδώ θα υποβάλω νέα προφορική τροπολογία ανάλογα με τις πληροφορίες που πήρα σήμερα το πρωί. Να διαγραφεί η μνήα στο συγκεκριμένο νόμο και να αναφέρονται οι τροπολογίες στην νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε η διατύπωση που βλέπετε εδώ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα λέμε ενθαρρύνει τις αρχές να υιοθετήσουν ρήτρες ασφάλεια σε όσον αφορά την νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης και να υπάρξουν επιπλέον διαβουλεύσεις και διάλογο σχετικά με τον νόμο αυτό, ώστε να υπάρξει ευρεία στήριξη από την δημοσιογραφική κοινότητα και τότε μόνο ο νόμος αυτός να περάσει. Αυτή είναι μια προφορική τροπολογία λοιπόν που θα υποβάλω βάσει των όσων έμαθα σήμερα. Για να είμαι σύντομο τώρα, δεν θα σας τα πω όλα. Για τη διαφθορά και την δικαστική υπηρεσία έχω δύο διαφορετικές παραγράφους. Ακολουθώ εδώ τις τροπολογίες Μακοβάη όσον αφορά τα κοινωνικά και την απασχόληση. Και προσπαθώ να φτιάξω ένα συνεκτικό κείμενο με τους κύριους Φαγιών και Φάρμ. Για τις γυναίκες Ξέρω ότι είναι ένα θέμα ευαίσθητο για το ΕΛΚ και άλλους συναδέρφους. Με ποιο τρόπο η νομοθεσία για την ε, παύση κοίησης πέρασε από το Κοινοβούλιο χωρίς προηγουμένως να γίνουν διαβουλεύσεις. Θέλω να είμαι σαφής ότι εγώ δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη μία ή την άλλη θέση, είναι ένα ευαίσθητο θέμα, το καταλαβαίνω αυτό. Πρόκειται για την κοινοβουλευτική διαδικασία που οδήγησε στο αποτέλεσμα που κατέληξε. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τον κατάλογο ψηφοφορίες και ελπίζω να μπορέσουμε τελικά να εγκρίνουμε τη δικιά μου τη διατύπωση και να μπορέσει και το ΕΛΚ να συμφωνήσει. Τελικά, πολλές τροπολογίες υπήρξαν στην έκθεση αυτή και πολλές από αυτές ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές. Θέλω να ευχαριστήσω και τους Έλληνες και τους Βουλγάρους συναδέλφους που ελπίζω να αισθάνονται ότι έχω συμπεριλάβει πολλές από τις δικές τους τροπολογίες χωρίς όμως το κείμενο ε, δυσανάλογα να αναφέρεται ε, σε συγκεκριμένες σχέσεις. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να με στηρίξετε στην τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα έχει κλείσει ο καταλόγος των αγορητών, 13 ομιλητές, ένα λεπτό καθένας. Κύριε Κούκαν, δεν μου διέφυγε το όνομά σας. Κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω το 1 και 25 δευτερόλεπτα, αν και είμαι σκέδος εισηγητής. Έχω αναφέρει επανειλημμένος ότι θέλω να είναι μια, η έκθεση αυτή ισορροπημένη, ώστε να δείχνει τη στήριξη και την αφοσίωσή μας στην ε, ένταξη της χώρας αυτής. Όμως θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά και τις πολιτικές και τις οικονομικές και τις οικονομικές εξελίξεις. Κατά την άποψή μου πρέπει να έχουμε επικοδομητική προσέγγιση ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους της Μακεδονίας να συνεχίσουν τη διαδικασία αυτή προς την ένταξη, όμως να τονίζουμε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή Χάουιτ, ο οποίος ακολούθησε αυτή τη γραμμή, όμως να ευχαριστήσω και του συναδέλφου για τι τροπολογίε του που συνεισφέρουν στο να γίνει η έκθεση ακριβέστερη. Νομίζω δεν θα ήταν δυνατόν να αποφύγουμε τελείω τι διαφωνίε σε απόψει όταν συζητούμε την έκθεση αυτή, ιδιαίτερα ε, όταν ε, συνομιλούμε με Έλληνε και Βουλγαρού συναδέλφου. Όμω προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καθησυχάσουμε και τι δικέ του τις ανησυχίες. Είχαμε καλή συζήτηση για τις συμβαστικές τροπολογίες. Καλωσορίζω εδώ την πολύ θετική ατμόσφαιρα που είχαμε σε όλε τι συναντήσει μας και νομίζω ότι ήταν πραγματικά μια συμπεριφορά κυρίων ε, και ε, μεγάλης ευγένειας αυτή που έδειξε ο εισηγητής μας. Καλωσορίζω την ε, έκκληση για έναρξη διαπραγματεύσεων με την ε, Μακεδονία καθώς και την ελληνική προεδρία να εκμεταλλευτεί το θετικό πνεύμα που υπάρχει σήμερα για να ξεφύγουμε από το τέλμα στις διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη ότι ως προς την ε, ένταξη της ε, Μακεδονίας εξετάζουμε και τα όρια της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην όλη διαδικασία ένταξης χωρών της περιοχής αυτής. Ε, θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι στάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου θα πρέπει να υλοποιηθούν και να δοθεί έμφαση σε αυτή, καθώς και η συμπελίωση των του κυβερνώντος κόμματος με την αντιπολίτευση θα πρέπει η παρακολούθηση των συνόρων επίσης να είναι ένα θέμα που θα ενταχθεί στη διαδικασία αυτή της προσχώρησης της χώρας. Να πω κάτι και στον εισηγητή. Ε, όταν λέτε για δίγλωση εκπαίδευση, σημαίνει ότι ένα μέρος του πληθυσμού θα πρέπει να μάθει τη γλώσσα του άλλου, τα αλβανικά. Εγώ είμαι στη Σλοβακία. Αν κάποιος μου λέγει ότι πρέπει να μάθω ουγγρικά, θα διαμαρτυρόμουν πολύ έντονα. Ρίτσαρντ, μήπως να το εξηγούσε καλύτερα. Ίσως εδώ να ήμασταν κάπως πιο ακριβείς στην αναφορά μας. Ευχαριστώ. Έτσι κι κρατήσατε την καλή σας εικόνα χάρη στην πρώτη σας παρέμβαση στην προηγούμενη συζήτηση. Κύριε Κορνέλισον. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Και πάλι μπράβο στον εισηγητή στον εισηγητή για μια που θα έλεγα ότι ασχολήθηκε με την πλέον πολιτικά ευαίσθητη έκθεση πρόοδου από όλε τι υπόλοιπε. Δύο παρατηρήσει. Ε, να υποστηρίξω τροπολογίε θέλω. Ε, πρώτα απ' όλα μια έκκληση στήριξη για την τροπολογία 53. Εδώ λέγεται ότι καλωσορίζει υπ' αυτήν την έννοια την πρόταση ενό σύνθετου ονόμου με γεωγραφικό προσδιορισμό όπω ο απεσταλμένο του ΟΗΕ έχει προτείνει και πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση για συμβαστική λύση λαμβάνοντα υπόψη την μακεδονία μακεδονική πολιτιστική ταυτότητα, ε, γλώσσα και ιστορία. Α εκμεταλλευτούμε αυτή την τροπολογία για να βρεθεί μια λύση ε, για τη Μακεδονία και να χρησιμοποιήσουμε τι περιορισμένε μα αρμοδιότητε ω κοινοβούλιο, αλλά για να κάνουμε μια σαφή και συγκεκριμένη δήλωση. Ελπίζω να κερδίσετε την πλειοψηφία η τροπολογία αυτή και Επίσης διερωτήθηκα πώς ε, σκοπεύει ο συγκεκριτής να επιλύσει τις διάφορες ε, τροπολογίες του κυρίου Γιάννη και δικές μας, την 1.41, 1.43, 1.63 και 1.67. Ε, τροπολογίες που αφορούν το πολύ σημαντικό ζήτημα για τα περιβαλλοντικά πρότυπα και την διαχείριση των υδάτων κυρίως. Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος ή ενεργειακής ε, διαχείρισης, από όσο επίσης υπάρχει μια σαφής απειλή εργοστασίων υδρογόνου που χτίζονται σε φυσικά, πολύ κοντά σε φυσικά πάρκα, σε προστατευόμενες περιοχές. Τι άποψη έχει ψυχητής για αυτά. Κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τα θερμότερα συγχαρητήριά μου προς τον συνάδελφο κύριο Χάουιτ και πάλι έχει κάνει μια πολύ καλή απόπειρα να καλύψει ένα από τα, όπως υπόθηκε, πλέον δύσκολα και προκλητικά ε, θέματα ε, της υποψήφιας αυτής χώρας που θα πρέπει να υπερβεί πολλά εμπόδια για να φτάσει στην έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενδεχόμενη ένταξή της. Η ομάδα πάντοτε στήριζε τις ευρωατλαντικές φιλοδοξίες της Μακεδονίας και ουδέποτε καταλάβαμε το θέμα της ονομασίας. Ελπίζουμε πραγματικά να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο και πραγματικά νομίζω ότι οι συμβαστικέ λύσεις που προτείνονται είναι μια πολύ καλή ε, κίνηση για να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο αυτό. Θα στηρίξουμε τις τροπολογίε που αφορούν τις βουλγαρικές αντιρρήσεις για τόσα συμβαίνουν στη Μακεδονία. Αλλά Έχουμε πολύ σοβαρή διαφωνία, έντονη διαφωνία σε σχέση με τη συμβαστική λύση 12. 12 για το θέμα του, της υποχρεωτικής δίγλωσης εκπαίδευσης. Θυμάμαι κάποια στιγμή πια ένα τσάι με τον πρόεδρο της Μακεδονίας και έλεγε ότι κατά την άποψή του η βασική γλώσσα των Δυτικών Βαλκανίων θα είναι τα αγγλικά ε, λίγο πολύ γλώσσα επικοινωνία. Τώρα, η ιδέα να επιβάλλουμε στους μένους να μάθουν τη γλώσσα των δε, νομίζω ότι είναι μια υπερβολή. Όπως υπόθηκε από τον κύριο Κούκαν, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στη Σλοβακία. Εκεί η επίσημη γλώσσα είναι τα σλοβακικά, αλλά κάποιες παραχώρησεις γίνονται για τις μειονοτικές γλώσσες, όπως τα ουγγρικά, και το ίδιο και με την ε, Μακεδονία, όπου η επίσημη γλώσσα είναι τα μακεδονικά, αλλά υπάρχει μία μειονοτική γλώσσα, τα αλβανικά. Νομίζω ότι πάμε πολύ μακριά ε, στο, σε μία διάθεση παρέμβασης, ε, ευρωπαϊκή προοπτική να μπούμε στα εσωτερικά, στι εσωτερικέ υποθέσει σε μια κυρίαρχη χώρα που έχει απόλυτη δικαιοδοσία για τέτοια θέματα στο δικό τη επικράτεια. Για την ε, τροπολογία λοιπόν 12 θα ήθελα να την ξαναδούμε και να σκεφτείτε αν ακριβώ εννοείται αυτό που λέει για την υποχρεωτική δίγλωση εκπαίδευση και την διδασκαλία αλβανικών σε όλου του Μακεδόνε και όλο τον πληθυσμό τη χώρα. Επίση να πω ότι έχω σοβαρέ συντηρήσει. Έχετε ξεπεράσει το κατά ένα λεπτό το χρόνο σα. Με συγχωρείτε, αλλά η άμβλωση δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να εμεί. Με Μπορείτε, λέει ο Πρόεδρος, να ακολουθήσετε τις ε, ε του Πρόεδρου, παρακαλώ. Σταματήστε. Ο κύριος δεν... Θα σταματήσουμε τώρα, γιατί άλλως δεν θα φτάσουμε... Δεν θα προλάβουμε όλα, όλα τα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ, παραμένετε πιστό στο ένα λεπτό. Δυόμιση λεπτά μιλήσατε, αντί για ένα. Κύριε Βούγεβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πλήρη και πλήρη καλών προθέσεων έκταση. Το πρόβλημα με τη Μακεδονία είναι ένα εμβληματικό παράδειγμα του πώς μπορούν να λυθούν τα προβλήματα αν υπάρχει καλή θέληση. Πρέπει εμείς να βοηθήσουμε να ξεπεράσει η Μακεδονία το θέμα της, ε, του ονόματος. Μήπως η ελληνική προεδρία δεν είναι η πιο εύστοχη χρονική στιγμή για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Κατά τα άλλα. Μια χώρα που έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και έχει δείξει μεγάλη θέληση για να κάνει μεταρρυθμίσεις θα τροχοπεδηθεί λόγω του θέματος του ονόματος. Και τι θα κάνει τότε. Θα στραφεί πάλι στο παρελθόν γιατί δεν έχει καμία άλλη επιλογή. Αν θέλουμε η χώρα αυτή να στραφεί προς το μέλλον θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και ιδιαίτερα η ελληνική προεδρία θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο γι' αυτό. Είναι απαραίτητες οι καλέ σχέσεις με τους γειτονές της. Λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης της Μακεδονίας ξέρουμε που είναι, ότι είναι <clears throat> περιστοιχιζόμενη από ποιες χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσει τις καλύτερες σχέσεις με τους γείτονές της και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή μας θα πρέπει να τους βοηθήσει. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, μετά από ένα λεπτό θα σας σταματάω αυτομάτως, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γεια. Κύριος Σαλαβράκος. Να είστε καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, uh, ο συγκητής κράτησε περισσότερο, λέει ο κύριο Στάνουκ. Εσείς πήλησατε πιο πολύ από όλου, ε, παρατηρεί ο πρόεδρο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως και αν εγώ συνέτασα μια έκθεση για τα Φόκλαντ θα εθωρούσα ανόητο το ότι έκανε πόλεμο η Μεγάλη Βρετανία για τα Φόκλαντ. Το ίδιο και ορισμένοι Εγγλέζοι θεωρούν για το όνομα της Μακεδονίας. Οι Έλληνες είναι τόσο ανόητοι όσο ανόητοι ήταν οι Άγγλοι που έκαναν πόλεμο για τα Φόκλαντ. Δεν έχουν αντιληφθεί το εξή ότι 20 χρόνια είναι αυτό το κράτος, έχουν περάσει 8 ελληνικές κυβερνήσεις και εκεί υπάρχει η κυβέρνηση μόνο ενός κόμματος η οποία επιμένει σε ένα όνομα καθαρά ελληνικό. Δεν έχει αντιληφθεί το εξής ίσως η ομάδα μας εδώ, ότι το κράτος αυτό διοικείται από τέος Έλληνες, τέος Έλληνες κομμουνιστές, οι οποίοι έφυγαν, έκαναν πεδομάζουμε από την Ελλάδα και πάνε και το κυβερνάνε τώρα και θέλουν την Ελλάδα, θέλουν τη Θεσσαλονίκη και δεν το έχετε αντιληφθεί. Πάτε να κάνετε προβλήματα σε μια χώρα που δεν υπάρχουν. Λοιπόν, επιμένω, όσο ανόητοι ήταν οι Εγγλέζοι που κάναν τα Φόκλαν, όλε μου τόσο ανόητοι είναι και οι Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, ε, είναι, είναι συνήθις νονή, ε, η συνήθις νονή και οι πολύ έξυπνοι αυτοί κύριοι οι οποίοι έχουν την καλύτερη άποψη για το... Σταματήστε παρακαλώ λέει ο πρόεδρος. Προκλήθηκε κύριε πρόεδρε. Από τον κύριο εδώ. Naravno, za osobito je još jedno odgađanje početka pre... Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Πίκουλα. Είναι λυπηρή η έλλειψη πρόοδου στις διαπραγματεύσεις με την Μακεδονία. Υπάρχουν όμως και μερικά θετικά στοιχεία, τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τα προβλήματα με την υποψηφιότητα της Μακεδονίας και να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της διαφθοράς. Θα πρέπει να είναι πιο διάφανα τα οικονομικά των κομμάτων και οι σχέσεις των πολιτικών με τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να σέβεται την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και όλα τα θέματα που υπάρχουν στη διοικητική δομή της χώρας αυτής. Αλλά η έκθεση προόδου δείχνει ότι ο λαός της Μακεδονίας είναι έτοιμος να προχωρήσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε θετικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Ρίτσαρτ, ευχαριστούμε πολύ για τις προσπαθίες σου. Καταλαβαίνουμε την ε, απογοήτευση πολλών Μακεδόνων πολιτών που δεν υπάρχει καμία πρόοδος ε, ως προς την έναρξη των διπλωματεύσεων ένταξης, όμως απογοήτευση θα υπάρξει και από τις μακεδονικές αρχές όταν ε, θα έπρεπε να υπάρχει μάλλον όταν διαβάζουν τις συστάσεις μας επιλεκτικά τα τελευταία χρόνια για σχέσεις καλής γειτονίας. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μόνο μία παρατήρηση γιατί δεν έχω και τόσο χρόνο για την ημερή συμφωνία μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων η οποία πρόκειται να υπογραφεί. Υπάρχουν δύο ε, σημεία, δύο σημεία που μας δυσκολεύουν. Πρώτα απ' όλα ότι η κυβέρνηση της Μακεδονίας δεν θέλει η δήλωση του 1999 για, τη συνταγματική για την παράγραφο του συντάγματος 49 ε, και που αναφέρεται στις σχέσεις Μακεδονίας και ε, Βουλγαρίας δεν θέλει να ε, συμπεριληφθεί και επίσης δεν θέλει η κυβέρνηση της Μακεδονίας να ακολουθήσει τις συστάσεις αυτού του σώματος για την καλύτερη συνεργασία και τις καλές, σχέση καλής γειτονίας με τις γειτονές χώρες. Ευχαριστούμε κύριο Στίαρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το βασικό μήνυμα αυτού του ψηφίσματο είναι ότι η Μακεδονία, όσο το θέλουν συντομότερα, θα πρέπει να περάσει σε διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα τη ονομασία. Όμω αυτό δεν είναι μέρο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων. Ε, εάν θέλουμε να αξιοποιήσουμε την συμμετοχή μα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιλύσουμε διμερεί προβλήματα, τότε το ευρωπαϊκό ιδεώδε δεν θα λάβει ποτέ σάρκα και οστά. Θα, θα ήθελα λοιπόν εδώ να στηρίξω την άποψη του κ. Κούκαν σε ό,τι αφορά το θέμα της δίγλωσης εκπαίδευσης και των δύο γλωσσών. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ακριβεί στην ε, αναφορά μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. και εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ για την έκθεσή του. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Στία. Κατά τη δική μας άποψη η Μακεδονία ήταν εταίρος μας στη διαδικασία προσχώρησης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς έχουμε υποστηρίξει την πορεία της. Δεν πρέπει να περνάει ο χρόνος και να μην λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη συνομιλιών. Με κάθε σεβασμό προς την ελληνική Προεδρία έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα η ένταξη της Κροατίας και θα πρέπει να βοηθήσει και την Μακεδονία τώρα. Μετά από την ένταξη λοιπόν <clears throat> αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από την διάσκεψη της Θεσσαλονίκη. Το θέμα του ονόματος δεν θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι για τις διαπραγματεύσεις και μόνο με τη συνέχιση των συνομιλίων μπορούμε να έχουμε πρόοδο στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να επενέσω τον κύριο Χάουτ για την πολύ καλή έκθεσή του. Γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και βλέπουμε ότι η πρόοδος έχει κάπως επιβραδυνθεί. Κατανοώ ότι κάποιες ε, προτάσεις μπορούν να συμπεριληφθούν στις συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό θα ήταν μια καλή λύση. Υπάρχει όμως μια προφορική τροπολογία που έχει κρατήσει την προσοχή μου, η τροπολογία 7. Θέλω να τονίσω εκεί το ότι υπάρχει ένα παρόμοιο κείμενο το οποίο έχει προταθεί. Ελπίζω ότι θα υποστηριχθεί. Όλα αυτά σημαίνουν την μελλοντική υποστήριξη Βουλγαρίας εναντί της Μακεδονίας. Κύριε Γιαννάκο. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή. Έκανε πραγματικά πολλές προσπάθειες, παρότι διαφωνώ σε ορισμένα σημεία μαζί του, ε, διείδα την προσπάθειά του να συγκεράσει τις απόψεις. Ε, θέλω να σημειώσω ότι δεν γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια από την πλευρά της χώρας αυτής και της κυβέρνησής της για να, λυθούν, για να λυθεί το θέμα του ονόματος. Το θέμα του ονόματος δεν είναι τυπικό. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Είμαστε 75 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και νομίζω ότι ξεχνάμε γιατί αυτός έγινε. Πληροφορήθηκα κύριε Πρόεδρε ότι αυτή τη στιγμή έχουν εκτυπώσει καινούργια χαρτονομίσματα με την κεφαλή του Αλεξάνδρου και διάφορα άλλα σύμβολα. Είναι φανερό ότι όχι μόνο δεν θέλουν, αλλά συνεχώς δημιουργούν και νέα προσκόμματα. Καλό τον εισηγητή να κάνει προφορική τροπολογία αυτός, εφόσον αυτό μέχρι αύριο επιβεβαιωθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Schön. Aber da müssen Sie keine Sorgen machen, die Münzen mit dem Kopf von Alexander sind seit 2400 Jahren nicht mehr gültig. Μα νομίζω ότι <laughs> μπορούμε να έχουμε μια τροπολογία που να λέει ότι δεν θα ισχύουν πια τα χαρτονομίσματα με το, την πρωτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κύριε Μπριζάγκητς. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Μπιτικόφερ. Wahrscheinlich in Württemberg. Ibrisagic. Σαν να είμαστε στη λέει ο πρόεδρος. Κυρία Μπριζάγκητς. Και εγώ. Και εγώ πηγαίνω προς την ίδια γραμμή, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι με ενδιαφέρει το θέμα των δύο γλωσσών. Εντάξει, καταλαβαίνω εσείς αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι θέλετε οι άνθρωποι που μένουν σε ένα χώρο να γνωρίζουν ένα στη γλώσσα του άλλου. Εντάξει, αυτό έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε αυτή την επιλογή, όπως στην Σλοβακία να είσαι υποχρεωμένο να μάθεις ουγγρικά. Μπορείς να ενθαρρύνεις, ας πούμε, στη Σουηδία τα φιλαδικά. Ναι, αλλά δεν θέλω να με υποχρεώνει κάποιος. Οπότε αντιλαμβάνομαι εδώ το κινητρό σας, αλλά πρέπει να αλλάξει πιστεύω η διατύπωση. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω τι εννοείται εδώ με τον όρο ultra-nationalism. Στην Σουηδία ξέρω ποιον θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε υπερεθνικιστή, αλλά σε αυτή την περίπτωση σε ποιον αναφέρεστε. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Αυτό το σχέδιο του εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση με την τέτοια Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη ε, Ιουγκοσλαβία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξέρετε ότι συνεχίζει να βοηθάει τη χώρα μέσω διαρθρωμένου διαλόγου και με, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ε, προχωρούν στις ε, προσαρμογές τους για να καλύψουν διάφορα κενά και να πλησιάσουν στις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διάφορες ανησυχίες πάντως όσον αφορά τις, την εφαρμογή συστάσεων για τον εκλογικό νόμο, για παράδειγμα. Όπως ε, είπε και ο συγκητής, γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει εξελίξεις τις τελευταίες εβδομάδες. Πρώτα απ' όλα εγκρίθηκε η νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης και τώρα περιμένουμε να δούμε ποιε είναι οι τροπολογίε που έχουν ε, κατατεθεί για τον νόμο αυτό. Επίση, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η διαβούλευση και προσαρμογή στις διεθνείς προδιαγραφές. Πάντα για τα μέσα ενημέρωσης που αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στην περσινή μας έκθεση πρόοδου, εδώ θέλουμε να συνεχιστεί ο διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δημοσιογράφους, ώστε να λυθούν και άλλα ζητήματα που προκύπτουν στον τομέα της δημοσιογραφίας. Έπειτα, για τον εκλογικό νόμο, πιστεύουμε ότι η διακομματική συμφωνία έχει οδηγήσει σε προτινόμενες αλλαγές και η συζήτηση γίνεται τώρα στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε οι αλλαγές αυτές όταν θα έχουν εγκριθεί θα βοηθήσουν να αντιμετωπιστούν διάφορα ε, θέματα που έχουν να κάνουν και με τις συστάσεις. Και έτσι θα διευθετηθεί το θέμα σχέσεων ε, κράτους και μέσων ενημέρωσης. Ο ο αξιότιμος κύριος Χόβιτ έχει κάνει διάφορες συστάσεις που θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάθος. Πάντως να ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγάλη σημασία σε μια κοινωνία των πολιτών που να είναι ενεργός και την στηρίζουμε. Θέλουμε όντως η κοινωνία των πολιτών να αποτελείται από διάφορα τμήματα του πληθυσμού της χώρας. Όπως ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για να αξιολογεί την έκθεση πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σα, τα οποία παίρνω πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, ήδη από την αρχή νομίζω ότι ήμουν πολύ σαφής. για την επιβολή. Εδώ λέμε προώθηση, δεν λέμε επιβολή, λέμε προώθηση της διγλωσίας και εκεί όπου υπάρχει πλειοψηφία άλλης γλωσσικής ε, γλωσσικού τμήματος κτλ. Λοιπόν, όταν λέμε promoting σημαίνει να προωθήσουμε, δεν σημαίνει να επιβάλλουμε και στη συμβαστική συνάντηση που είχαμε κανένας δεν είχε αντίρρηση δεν υπήρχε πρόθεση επιβολής κανένας από τους σκιώδεις δεν σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Και αυτή είναι η δημοκρατία. Αν κάποιο είχε αντίρρηση, έπρεπε να το έχει πει. Ή αν κάποιο αισθάνεται ότι η ερμηνεία είναι άλλη από αυτή που θέλουμε, ευχαρίστω θα προσπαθούσα να το αλλάξω. Αλλά όπω είπε και ο κύριο Κόκαν και άλλοι, αν έχετε κάποια καλύτερη πρόταση, ελάτε να μου την πείτε. Πάντως πρόθεσή μας δεν ήταν υποχρεωτικά να επιβάλλουμε δύο γλώσσες. Και δεν θα ήταν και ρεαλιστικό. Για τον όρο ultra-nationalism. λέει ότι καταδικάζει κάθε είδους υπερεθνικισμό στη χώρα. σε, σε, σε κάποια χώρα, in a country, δεν μιλάει για συγκεκριμένη χώρα, Λέει in a country. Σε μια χώρα. Αν βάζαμε εθνικισμός θα ήταν χειρότερο. Γιατί τότε θα στέλναμε το μήνυμα σε όλες αυτές τις χώρες που θέλουν να ενταχθούν. Γιατί, όπως είπα και πριν, ο εθνικισμός μερικές φορές βερβεύεται με τον πατριωτισμό. Αλλά επειδή ακριβώς έβαλα το ούλτρα, Νομίζω ότι φαίνεται πως δεν κατηγορούμε κανέναν στη χώρα τη συγκεκριμένη για ουλτραεθνικισμό. Λέει a «Ε, country, δεν λέει αυτή η χώρα. Δεν λέει στην χώρα, λέει σε μια χώρα. Για τα υπόλοιπα, κύριε Κορνέλισον, το 53 και για τη γεωγραφική διάσταση εδώ εγώ αντιστάθηκα τα προηγούμενα χρόνια και πάλι θα βάλω κατά συνείδηση ψήφο. Καλά, να πάω πιο γρήγορα, λέει ο κύριος Χόβιτ. Οι πράσινοι μου ζήτησαν τη γνώμη μου για το 1.41.43.166. Πρώτα απ' όλα, οι βούλγαροι συνάδελφοι ξέρω ότι είναι έτοιμοι για συμβιβασμό και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να καταλήξουμε σε ένα σεβασμό ώστε να αντεκατοπτρίζονται εδώ οι δικές τους ιδέες. Για τον κύριο Κόβατσοφ, δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα γιατί έχω καθίσει με τις αρχές της χώρας, το έχουμε δει, το έχουμε συζητήσει. Αλλά όσον αφορά τις κοινέ ε, εκδηλώσεις για κοινέ επαιτίου, συμφωνώ. Για, τον κύριο, για την κυρία Λουτσέβιτς ευχαριστώ να συζητήσουμε μετά διμερώς. Ευχαριστώ για την υπομονή σας, Πρόεδρε. Όπως καταλαβαίνετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η χώρα και η έκθεση αυτή. Η επόμενη έκθεση θα κάνει με την Ινδονησία, με την Άννα κατά πρώτον να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτριες ε, για την συνεργασία τους, την κυρία Ομερόιτεν, τον κύριο Βότσον, τον κύριο Μπουτιγκόφερ, τον κύριο Σόλτς. Ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική και επί της ουσίας η συνεισφορά τους. Και έτσι ενισχύθηκε η έκθεση αυτή. Η Ινδονησία είναι μια άκρο σημαντική χώρα. Πολύ και θα πρέπει πραγματικά να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδονησίας, Θα θεωρούμε στρατηγικές. Η Ινδονησία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παρουσία μουσουλμάνων στον κόσμο, είναι δημοκρατική χώρα, είναι μέλος του G20, είναι ιδρυτικό μέλος της ASEAN, είναι μέρος ε, της, ε, του τη διάσκεψη των μουσουλμανικών κρατών και δεν νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει μεγαλύτερη πολιτική και στρατηγική εμπλοκή στις σχέσεις της με την Ινδονησία. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια ανθεί η συνεργασία των δύο περιοχών αυτών του κόσμου, αλλά όχι σε πολιτικό επίπεδο. Η έκθεση αυτή όμως ε, ακριβώς ασχολείται με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας η οποία υπεγράφει το 2009, τελικά υπεγράφει από όλα τα 29 κρατημέλη από τα 28 κράτη-μέλη, οπότε είναι σημαντικό πλέον το Κοινοβούλιο να δώσει μια νέα όθηση στην συμφωνία αυτή. Υπάρχει μεγάλο πεδίο ανάπτυξης ε, των σχέσεών μας με την Ινδονησία σε όλα τα επίπεδα, από το οικονομικό και πολιτικό μέχρι ε, το κοινωνικό που έχουμε κοινέ προκλήσεις. Δεν πρέπει να παραμελούμε βεβαίως και την πτυχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, καθώς και τις καλή κυβέρνηση του κράτους δικαίου. Αυτά μπορούν να βελτιωθούν και οφείλουν να βελτιωθούν στην Ινδονησία. Αν και υπάρχει ήδη σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Πάντω βλέπουμε ακόμη κάποια πολύ αρνητικά στοιχεία να συνεχίζονται και να υπάρχουν. Λόγου χάρη ότι υπάρχει υποχρεωτική διδασκαλία θρησκευτικών, μουσουλμανικών μαθημάτων εις βάρος άλλων θρησκευτικών πεπιθήσεων, διότι η Ινδονησία είναι μια χώρα με τεράστια ποικιλία. Υπό όλες τις έννοιες, ακόμη και στο, στη θρησκευτικά πιστεύω των πολιτών της. Αλλά δεν μιλούμε μόνο για οικονομικούς χώρους, αλλά για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Εκεί κάποια πολλαπλά προβλήματα δεν έχουν ε, αντιμετωπιστεί, λόγω χάρη με τις δασικές πυρκαγιές, την ε, παράνομη υλοτομία, αλλά και άλλους τομείς όπου η συνεργασία θα μπορούσε να ενταθεί και προς όφελος δικός μας, δικό μας και της Ινδονησίας. Λόγου χάρη η ναυτιλιακή συνεργασία. Αλλά και ό,τι έχει να κάνει με την ε, φορολογία, ή ε, το κράτο δικαίου, ή την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Αυτό είναι κάτι που αφορά και θα έπρεπε να ανησυχεί την Ινδονησία. Και θα έπρεπε να μας απασχολεί και εμά, Διότι η ανταλλαγή εμπειριών θα ήταν πολύ αποτελεσματική. Σημειώνουμε επίση πολλέ πτυχέ ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίω των γυναικών. πτυχές που αφορούν τις προσπάθειες ε, ριζοσπαστικών ομάδων να προσπαθήσουν να ε, εγκατασταθούν και να ριζώσουν και στην Ινδονησία. Πράγμα που έχει συνέπειες ως προς την διακριτική μεταχείριση και την παρενόχληση πολλών πληθυσμικών ομάδων. Ομάδες όπως η ομάδα Αχμαντία. Το θέμα των ανθρωπίνων λοιπόν δικαιωμάτων είναι ένα ε, ζήτημα που έχει να κάνει και με οικονομικές και με κοινωνικές πτυχές όπως με τους Παππούα ε, που θα έπρεπε να μπορούν να επωφελούνται από τους πόρους της περιοχής τους ως ε, νόμος πληθυσμός της χώρας αλλά επίσης ξέρουμε ότι η αντιπροσωπεία μας οργανώνει μια ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή των Παππού αυτή την εβδομάδα. Αυτό μας απασχολεί λόγω των προσφάτων εξέλιξεων και επειδή θα έχουμε τώρα τον πρόεδρο του Ινδονησιακού Κοινοβουλίου και θα συνεντεθούμε μαζί του και εγώ με τους σκιώδεις εισηγητές και όταν μας άκουσε πραγματικά έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο να συνεργαστούμε και να καταγράψουμε τα προβλήματα που ακόμη αντιμετωπίζει η Ινδονησία στην Παπούα. Και αυτό σε ένα πνεύμα συνεργασίας, όπως ήδη έδειξε η Ινδονησία στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση των προβλημάτων που είχε με τους Άτσε. Εδώ λοιπόν θα έχουμε και άλλες συζητήσεις με τους πιο εισηγητές γιατί κάποια ζητήματα ακόμη πρέπει να επιληθούν και με τους πρασίνους. Νομίζω έχουμε 18 τροπολογίες αλλά φαντάζομαι ότι θα τα καταφέρουμε και ότι θα είναι απλή ψηφοφορία για όλους. Ευχαριστώ. Χρόνος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οι Αναγκόμες πολύ σωστά υπογράμμισε τις αλλαγές που έχουν λάβει η χώρα στην Ινδονησία, αλλά και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είναι τα θέματα της διαφθοράς, η προστασία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των μειονοτήτων. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεσή της, γιατί χαιρετίζει εξάλλου και τις πάρα πολύ θετικέ εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα στην Ινδονησία μετά από την πτώση του καθεστώτος Σουχάρτο το 1998. Στα τελευταία αυτά 15 χρόνια η Ινδονησία έχει κάνει ουσιαστική πρόοδο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρασία και το κράτο δικαίου. Έχει αναπτύξει μια ισχυρή οικονομία και σωστά αντιμετωπίζεται σαν μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ΑΣΕΑΝ. Η θέση αυτή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικροτεί αυτές τις εξελίξεις και εξασφαλίζει και μία εξισορροπημένη στάση έναντι της Ινδονησιακής κυβέρνησης. Πιστεύουμε ότι οι ε, εναπομένουσες <clears throat> προκλήσεις θα αντιμετωπιστούν και τονίζουμε την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας για να μπορέσουμε να εδραιώσουμε μια καλή εταιρική σχέση με την ε, Ινδονησία. Για τον κατάλογο ψηφοφορίας έχω ορισμένα προβλήματα. Δέχτηκα ορισμένε από τις τροπολογίες σας και εσείς ορισμένε από τις δικές μου αλλά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις στον κατάλογο ψυχοφορίας που θα πρέπει να τροποποιηθούν. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες όπου εγώ δεν έχω μεν αντίρρηση, αλλά αν δεχτεί κανείς όλες αυτές τις τροπολογίες θα έχετε μια τεράστια έκθεση και επίσης και περιπτώσεις που είναι αντιφατικά αυτά τα οποία λέγονται, άλλοτε λέτε υπέρ της ανάπτυξης και άλλοτε κατά της ανάπτυξης. Ίσως λοιπόν με τον κύριο Βάτσον και μαζί σας θα μπορούσαμε να βραχύνουμε λιγάκι αυτή την έκθεση και να βρούμε τα σημεία όπου υπάρχουν κάποιες αναντιστοιχίες. Ευχαριστώ. Λέω πρώτος χωρίς μικρόφωνο πάντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κύριος Μπιτικόφερ. Θέλω να συγχαρώ την κυρία Γκάμες για την έκθεσή της και θέλω επίσης να την ευχαριστήσω και για το ότι προσπάθησε να συμπεριλάβει όλα όσα είπαν οι σκιώδεις όλα όσα συμπεριλαμβάνουν οι διάφορες τροπολογίες και να τις συμπτύξει σε συμβαστικές. Είχαμε τέσσερις και χαίρομαι που βλέπω επίσης ότι στον κατάλογο ψηφοφορίας λαμβάνονται υπόψη δικές μας επιθυμίες. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά να θίξω ένα πρόβλημα ή ενδυνάμει πρόβλημα, δυνητικά, που βλέπω με την συμβιβαστική τροπολογία 11. Έχει δουλευτεί βέβαια η γλώσσα, αλλά εξακολουθεί να λέει, και βέβαια δεν το έχω ακριβώς εδώ, αλλά λέει ότι με θλίψη διαπιστώνει ότι όλο και περισσότερο Ισλαμική διδασκαλία συμμετέχει στην ε, εκπαίδευση και ότι αυτό μπορεί να είναι αιτία για την ανερχόμενη βία κλπ. Για μένα η διατύπωση αυτή είναι προβληματική. Τι θα πει οδηγεί στην αύξηση επεισοδίων. Πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατό αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε συμβάλλει. Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε μια διαφορετική διατύπωση. Η διατύπωση αυτή φοβάμαι ότι δεν βοηθάει. Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διατύπωση, θα βρεθούμε σε πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο σκιώδης ηγητής μας, Γκραμ, μου ζήτησε να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία μεταξύ της εισηγήτριας και των σχεδόν εισηγητών. Εκείνο υπογραμμίζει ότι η προσπάθεια που έγινε για τις συμβαστικές τροπολογίες οδήγησε σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Θέλει να υπογραμμίσει ότι οι περισσότερες επενδύσεις και εμπόριο με την Ινδονησία είναι αυτό που χρειάζεται και προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνανε και διάφορες τροπολογίες οι οποίες ε, υποβλήθηκαν ότι χρειάζεται επίσης περισσότερη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και οι τροπολογίες αυτές αναφέρουν επίσης την ανάγκη για παρετέρω συνομιλίες όσον αφορά τις θεωρήσεις. Επίσης πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθούν ε, οι ανταλλαγές μεταξύ των ανθρώπων μέσω του Erasmus Mundus για παράδειγμα, ή να οργανωθούν σεμινάρια ώστε να υπάρξει πιο στενή συνεργασία μεταξύ όλων των πλευρών. Είναι επίσης σημαντικό ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδονησίας να ενισχυθεί. Ο κύριος Graham έχει ακριβώς υποβάλει τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση που ελπίζει να στηρίξουν οι συνάδελφοι. Τονίζει επίσης ότι ελπίζει οι συνάδελφοι να εγκρίνουν την τροπολογία 52, να τη στηρίξουν δηλαδή, που αναφέρεται στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Όσον αφορά θανατική ποινή. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα καταφέρουμε μέχρι αύριο να καλύψουμε τις παρατηρήσεις που έγιναν και από τη Ρία και από τον κύριο Μπουτικόφερ. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι προτάσεις που θα μπορούσαν να διατυπωθούν πιο θετικά, πιο επικοδομητικά. Κατανοώ αυτά που ανέφερε η Ρία σε σχέση με τις παρατηρήσεις του κυρίου Βότσον δεν έχουν καλυφθεί από τις συμβαστικές τροπολογίες. Κάποιες φορές υπάρχουν εμνίες μεν, αλλά όχι ακριβώς με την ίδια διατύπωση του κυρίου Βότσον. Θα τα διατρέξω και πάλι. Και φυσικά δεν θα παραβλέψω τις συνεισφορές του κυρίου Βότσον, ακόμη και αν υπάρχουν στοιχεία που είναι κοινά με τις συμβαστικές, αλλά όντως μπορεί να βρούμε κάποιο τρόπο να συνδυάσουμε τις διατυπώσεις. ιδίω σε ένα σημείο νομίζω ότι είναι ευαίσθητη η γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουμε όταν μιλούμε για απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Εάν, ε, ακόμη και αν αυτό γίνεται με μια πολύ διορατική προσέγγιση στα πράγματα, διότι λέει start looking at negotiations, να αρχίσει να ε, στρέφει το βλέμμα προς Νομίζω ότι αν βρίσκαμε κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Και πάλι να ευχαριστήσω τους πάντες. Ο κύριος Βότσον πραγματικά έκανε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και επί της ουσίας συνεισφορές που, για θέματα που ξέρω ότι τον ενδιαφέρουν και είναι πολύ σημαντικά για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας. Γνωρίζω καλά την Ινδονησία. Έχω πάει πολλές φορές, πρέπει να πω ότι την αγαπάω τη χώρα αυτή και ξέρω ότι μας κοιτάνε με μεγάλη προσοχή από τη χώρα εκείνη, εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ινδονησία έχει κάποιους ιδιαίτερους δεσμούς με χώρες όπως η Ολλανδία, οι κάτω χώρες. Πραγματικά τους εκπλήσει πώς εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γνωρίζουμε τόσο πολύ και συνεχίζουμε να γνώμε την Ινδονησία. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να αρχίσουν να μετακινούνται και να ενταθεί και η συνεργασία μας ε, σε όλα τα επίπεδα. Δυστυχώ θα πρέπει να διακόψουμε λιγάκι την συζήτηση γιατί ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι πρώτον θυρών μας. Κύριε Τάνο, και ίσως θα πρέπει να επανέλθουμε σε κάποια άλλη ευκαιρία. Επαναλαμβάνει στα αγγλικά ο πρόεδρος ότι ο πρόεδρος Συμβουλίου είναι εδώ ήδη, οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να καλωσορίσω ένθερμα τον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, τον κύριο Βενιζέλο. Χαίρομαι για την παρουσία του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για πρώτη φορά και χαίρομαι επίσης για την ε, προσδοκόμενη συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία και τον κύριο Βενιζέλο Είχαμε ήδη πριν από δύο εβδομάδες την ευκαιρία να συναντηθούμε μαζί του στην Αθήνα. Και έχουμε φυσικά πιστεύω πάρα πολλούς λόγους για να συνεργαστούμε και είμαστε απόλυτα έτοιμοι από τη δική μας πλευρά. Κύριε Βενισέλο, θέλετε να μας παρουσιάσετε και τα, α, τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, αλλά φυσικά και τα συμπεράσματα του, Συμβουλίου, τα θέματα αυτά θα πρέπει να είναι και αλληλένδετα εξάλλου. Θέλω να χαιρετήσω επίσης και τον κύριο Πρεσβευτή της Ελλάδος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μια επιτροπή πολύ υψηλού κύρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι προτεραιότητε τη ελληνική προεδρία του εξαμήνου αυτού στα θέματα τη αρμοδιότητα τη περιοδική προεδρία, δηλαδή κυρίω στα θέματα τη διεύρυνση, αλλά με την ευκαιρία πριν από αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να παρουσιάσω εκ μέρου τη υπάτη εκπροσώπου τη κυρία Άστον τα σημεία της σημερινή συζήτησή μα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων It's a great pleasure for me to report to the Foreign Affairs Committee on the main points considered at the foreign... Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να σας μεταφέρω τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που έλαβε χώρα σήμερα. Προείδρευε η είπατε εκπρόσωπο, η Κάθριν Άστον, ήταν ο Επίτροπο Φίλου που είναι υπεύθυνο για τη διεύρυνση, ο Επίτροπο Μπίρκαλ υπεύθυνο για την ανάπτυξη και η Επίτροπο Γεωργίευε υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια επειδή συζητήθηκαν διάφορα θέματα που τους αφορούν στο σημερινό Συμβούλιο. Είπα εκπρόσωπος λοιπόν ξεκίνησε υπενθυμίζοντας τα θύματα της βομβερδιστικής επίθεσης στην Καμπούλ, όπου έχασαν τη ζωή τόσοι άνθρωποι και αναφέρθηκε και στους ε, θανάτους και των ε, υπαλλήλων το ΙΕ και άλλων εξωματούχων. Το θέμα, ένα βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν οι σχέσεις με τις γείτονες χώρες. Αναφέρθηκε στην σύραξη λοιπόν στη Συρία και τις επιπτώσεις στις γείτονες χώρες Λίβανο και και υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει στήριξη στη συνομιλίες της Γενέβης 2. Αναφέρθηκε επίσης τον κύριο Μπραχήμ που είναι εκπρόσωπος και αναφέρθηκε στην ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια και στην ε, διάσκεψη στο κουβέρτι 15 Ιανουαρίου. Η υπογράμμιση ότι είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των γυναικών στην ερνευτική διαδικασία και από σε φόρο τιμή στι προσπάθειε τη Ολλανδία και για τη συμμετοχή των γυναικών, λέγοντα ότι η φωνή των γυναικών μπορεί να βοηθήσει οι προτεραιότητέ μα να αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα τη ερνευτική διαδικασία. Πολλές χώρες ε, μέλη αναφέρθηκαν στην ε, πρόσκληση του Ιράν στη Γενέβη που οδηγεί σε κάποια βεβαιότητα κατά πόσο τελικά η πολίτευση της Συρίας θα συμμετέχει όχι. Επίσης αναφέρθηκε στο ρόλο των ε, διαφόρων πλευρών και χώρες μέλη υπογράμμισαν ότι όλες οι πλευρές που συμμετέχουν στις νομιλίες της Γενέβης πρέπει να δεχτούν τα αποτελέσματα και να, προηγουμένως να βασιστούν στις αποφάσεις του Ιουνίου του 2012 στο ανακοινωθέν τη ημερομηνία αυτή. Πρέπει να τονιστεί επίσης η ανθρωπιστική πτυχή τη κρίση έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά το οποίο υπογράμμισαν πολλοί υπουργοί. Είπατο εκπρόσωπο επίση εξέφερε τι ανησυχίε τη ότι η σύγκρουση αυτή μπορεί να έχει επιπτώσεις στις γείτονες χώρες, Λίβανο και Ιράκ, με βία που μπορεί να εξαπλωθεί. Τέλος, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμπεράσματα όσον αφορά τη Συρία. Το δεύτερο σημείο ήταν η Αίγυπτος η ύπατος εκπρόσωπος αντέδρασε στα αποτελέσματα του ε, δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα για το Σύνταγμα στις 14 και 15 Ιανουαρίου. Η ύπατος εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να υποστηρίζει τους Αιγύπτιους προκειμένου να πετύχουν τα όσα ζήτησαν με την επανάσταση του Ιανουαρίου του 2011. Αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ασφάλεια, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και καλύτερη οικονομία παραμένουν στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα επιτεύγματα της Αιγύπτου. Επίσης αναφέρθηκε σε νέο πολιτικό διάλογο εν ώψη δημοκρατικών αλλαγών μια σωστή εκπροσώπηση των διάφορων πολιτικών απόψεων στο μελλοντικό κοινοβούλιο, λογοδοσία της κυβέρνησης και των θεσμών και μεγαλύτερη ασφάλεια και βιβλία για όλους. Είπα της εκπρόσωπος εξέφρασε την ανησυχία της για την πρόσφατη βία και για την επιδείνωση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλές χώρες μέλη υπογράμμισαν τη σημασία που έχει η πολιτική σταθερότητα στην Αίγυπτο, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συμμετοχή όλων στη διαδικασία. Η παρουσία παρατηρητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τι κοινοβουλευτικέ και προεδρικέ εκλογέ στη χρονιά αυτή αναφέρθηκε επίση, όπω επίση και οι οικονομικέ προκλήσει που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος. Το τρίτο σημείο ήταν η ειρνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενημερώθηκε από τον ύπατο εκπρόσωπο για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την ειρνευτική αυτή διαδικασία. ΥΠΑΤΟ εκπρόσωπο επιβεβαίωσε ότι οι εργασίε συνεχίζονται για την εφαρμογή των συμπερισμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013. Θα θυμόσαστε ίσω ότι το Δεκέμβριο το Συμβούλιο εξέφρασε την πλήρη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι συνεχιζόμενε προσπάθειε των πλευρών και των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να υπάρξει ένας διακανονισμός για την σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Και το Συμβούλιο επίσης ε, προειδοποίησε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν ε, δράσεις οι οποίες να υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις αυτές. Επιπλέον επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει ουσιαστικά σε ε, διακανονισμούς και διευθετήσεις μετά την σύγκρουση αυτή για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Συμφωνίας Ειρήνης και ότι μπορούμε να περιμένουμε ένα τεράστιο πολιτικό, οικονομικό και ασφάλειας πακέτο από πλευρά στην Ευρώπη προς τις δύο πλευρές. Και προκειμένου να υπάρξει μια τελική ειρηνευτική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει και να βοηθήσει και το Ισραήλ και το μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης για να βρεθεί η λύση των δύο χωρών και να καταλήξουμε σε μια ειρήνη διαρκείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει λοιπόν και στις δύο πλευρές μια συνεργασία ειδική με πρόσβαση στις αγορές, ε, πιο στενές πολιτιστικές και επιστημονικές σχέσεις, αλλά και πρόθεση των σχέσεων των επιχειρήσεων μεταξύ τους. Όπως επίσης θα δοθεί όθηση σε πολιτικό διάλογο και σε συνεργασία για την ασφάλεια. Αφγανιστάν, το Συμβούλιο στέλνετε σε λυπητηριά τους τις οικογένειες των εξωματούχων που έχασαν τη ζωή τους και επαναλαμβάνει την ε, επιθυμία της Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει και να στηρίξει τα συμπεράσματα για την κατάσταση του Αφγανιστάν μετά το 2014. Επαναλαμβάνει την ε, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μακράς διάρκειας εταιρική σχέση με το Αφγανιστάν και ζητάει να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις όσον αφορά την ε, Συμφωνία Συνεργασίας και εταιρική Σχέσης μεταξύ Αφγανιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θέλει να δώσει τεχνική και οικονομική βοήθεια για να ενισχυθεί η εκλογική διαδικασία. Εξέφρασε επίσης την ανησυχία της όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και κατευθυντήριες ε, γραμμές για τη στρατηγική όσον αφορά το Αφγανιστάν θα υιοθετηθούν για να αντικαταστήσουν τις σημερινές κατευθυντήριες γραμμές μετά το 2016. Κατά τη διάρκεια του γεύματος συζητήθηκαν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγικούς εταίρους. Ρωσία, για παράδειγμα, η προετοιμασία της διάσκεψης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας που θα λάβει χώρες 28 Ιανουαρίου. Επίσης υπογραμμίστηκε εκεί η σημασία που έχουν ε, οι σχέσεις αυτές με την Ρωσία σε σχέση με τα, τις τελευταίες εξελίξεις, ιδιαίτερα τις εταιρικέ σχέσεις με τις ανατολικές χώρες, ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταλλάξαμε υπόψη επίσης για την σε εξελίξεις μετά τη διάσκεψη του Βίλνιους. Συζητήθηκε επίσης το... Προτάθηκε μάλλον να συζητηθεί παρετέρω η κατάσταση τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ουκρανία τώρα. Εκφράστηκαν ανησυχίες για τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της ε, Ουκρανίας την Πέμπτη που μας πέρασε, λέγοντας ότι ελήφθησαν με μη δημοκρατικό τρόπο και ότι πρόκειται για πολύ αμφιλεγόμενα ζητήματα. Επίσης αναφερθήκαμε στις διαμαρτυρίες στην πλατεία Μαϊντάν και είπαμε ότι κινδυνεύει να επιδεινωθεί η κρίση και να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στις αξίες της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Υπογραμμίσαμε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε πιο στενά το θέμα αυτό και να σταθμίσουμε τα μηνύματα τα οποία στέλνουμε. Υιοθετήσαμε συμπεράσματα λοιπόν για το σημείο αυτό. Και έρχομαι τώρα στο Ιράν είπα το εκπρόσωπο ενημέρωσε για την εφαρμογή του καινού σχεδίου δράσης ανάμεσα στο Ιράν και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συντρία. Και βάσει αυτού το Συμβουλίο ενέκρινε νομικές πράξεις για να άρει κάποιες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Πήραμε την έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας ότι ακολουθεί τις δεσμεύσεις του το Ιράν σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα δράσης. Οπότε με τους εταίρους μας συμφωνούμε με την έκθεση αυτή και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά αποφάσισε σήμερα το απόγευμα ότι άρουμε τα περιοριστικά μέτρα για τέσσερις πτυχές που έχουν να κάνουν με τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν για τις εξαγωγές ε, πετροχημικών, ε, πετρελαίου και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής. Σύμφωνα με το συμπέρασμα, το Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του Υπογραμμίζω την ιδιαίτερη συζητηγή κατάσταση στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. Το Συμβούλιο ενέκρινε συμφωνία για τις μελλοντικέ δράσεις ΚΕΠΑ και για την διαχείριση της κρίσης. Πολλές χώρες μέλη όμως πρέπει να έχουν την συμφωνία του κοινοβούλιο τους. Οι στρατιωτικές δραστηριότητε εκεί θα συνεισφέρουν να υπάρξει ένα ασφαλές και σίγουρο περιβάλλον και θα δώσουν προσωρινή στήριξη για να διασφαλιστεί πλήρως η ανάπτυξη της, ε, αποστολή, της αποστολής ε, εκεί, της ΑΦΣΙΜΚΑΡ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει προσωρινά στήριξη μέχρι έξι μήνες για να βοηθήσει να επιτευχθεί ένα ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή και μετά να αναλάβει η Αφρικανική Ένωση. Το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ιδιαίτερα την δυνατότητα η ΜΙΣΚΑ να συμμετάσχει σε ειρηνευτική αποστολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει για να προστατεύσει τον πληθυσμό που κινδυνεύει περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια που είναι ο μισός πληθυσμός ουσιαστικά της χώρας. Βάσει της απόφασης 19ης Δεκεμβρίου εκφράζει τη βαθιά ανησυχία για την κατάσταση, τη στήριξή του στην αφής καρ και στηρίζει την IFM CAR. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ήδη τις προσπάθειες σταθεροποίησης στην κεντρική Αφρική για να προστατευτούν οι πολίτες και να υπάρξει σταθεροποίηση στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει 50 εκατομμύρια ευρώ από την διευκόλυνση για την ειρήνη στην Αφρική για να στηρίξει την αποστολή της και η Μίκο Πάξ έχει πάρει 55 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κύριος ε, εταίρος ανθρωπιστικής βοήθειας και ανάπτυξης στην Κεντρική Αφρική με 2 από τα 4,6 εκατομμύρια Συνεισφέρει λοιπόν με την ανθρωπιστική βοήθεια και το 2013 η ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε στα 77 εκατομμύρια. Το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μία αερογέφυρα για να μεταφέρει αγαθά και τρόφιμα στη χώρα. Τέλος, Νότιο Σουδάν. Συζήτηση έγινε για την σοβαρή κρίση στο Νότιο Σουδάν. Από τότε που ξέσπασε η κρίση το Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε έκκληση για σάμεση κατάπαυση του πυρός και ζήτησε διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση ειρηνικά και δημοκρατικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις προσπάθειες δεμεσαλόβησης της διακυβερνητικής αρχής για την ανάπτυξη. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου όσον αφορά τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τώρα μπορώ να συνεχίσω στα ελληνικά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας. Είχαμε την ευκαιρία στη συνάντησή μας με το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και με τους Προέδρους των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ιδίω κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Επιτροπής του κ. Μπρόκ στην Αθήνα, να παρουσιάσουμε αναλυτικά τις μεγάλες πολιτικές προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας. Οι προτεραιότητες αυτές είναι οι προτεραιότητες όλων των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Γιατί προφανώς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες αυτή τη στιγμή τους απασχολεί το ζήτημα της επανόδου σε θετικού ρυθμούς ανάπτυξης, το ζήτημα της ανεργίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους Ευρωπαίους πολίτες, το ζήτημα της διαφύλαξης της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου. Όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τους απασχολεί το ζήτημα της ενίσχυσης των θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης στο επίπεδο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του ευρώ. Με βασικό θέμα την περίοδο αυτή την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Όλους μας απασχολεί και ιδίως τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις μεσογειακές χώρες, το ζήτημα της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, το ζήτημα της κινητικότητας, η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η κατανομή των βαρών μεταξύ των συνοριακών και παράκτιων χωρών και όλων των άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές είναι και οι τρεις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας οι οποίες εξειδικεύονται στις επιμέρους συνθέσεις του Συμβουλίου. Η τέταρτη οριζόντια προτεραιότητά μας είναι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, ιδίω η μεσογειακή πολιτική που ξεκινά από την αλληλεία, φτάνει στο περιβάλλον, στην ποσοσία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καταλήγει στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών δεν μνημονεύεται ρητά ως προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας το ζήτημα της διεύρυνσης και ιδίως το ζήτημα της διεύρυνσης με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και αυτό γίνεται γιατί όπως γνωρίζετε η διεύρυνση και ιδίως η ευρωατλαντική και πιο συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων ήταν η πρώτη προτεραιότητα της προηγούμενης ελληνικής προεδρίας του 2003. Οι προηγούμενες ελληνικές προεδρίες ταυτίστηκαν με μεγάλα κύματα διεύρυνσης. Η Προεδρία του 1994 που κορυφώθηκε στο, στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας έχει σφραγίσει την μετάβαση από την Ευρώπη των 12 στην Ευρώπη των 15. Και κατά τη διάρκεια της, της τελευταίας Προεδρίας του 2003 είχαμε την τελετή ένταξης 10 νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υπογραφή της Συνθήκης των Αθηνών. Ιδίως η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων που ήταν το κύριο σημείο της Ατζέντα 2014 της προηγούμενης ελληνικής προεδρίας έχει πλέον υιοθετηθεί από το Συμβούλιο, είναι η τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική, άρα δεν αποτελεί πρόταση της σημερινής ελληνικής προεδρίας, γιατί η υποχρέωσή μας είναι να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που έχει ήδη πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά από την προετοιμασία που έγινε στο επίπεδο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιετούς προσπάθειας σε πολύ μεγάλο βαθμό αντανακλώνται στο γεγονός ότι αύριο πραγματοποιείται η διακυβερνητική διάσκεψη για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Σερβίας, κάτι που το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή προοπτική όχι μόνο της Σερβίας, αλλά και για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κωσόβου ενώ στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου αποτυπώνονται οι θέσεις του Συμβουλίου για όλες τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Για την Αλβανία, όπου η δική μας θέση ήταν πως θα έπρεπε από τώρα να παρασκευθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, αλλά αυτό θα το επανεξετάσουμε σύμφωνα με την κοινή μας θέση τον Ιούνιο. Περιλαμβάνεται η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με το Μαυροβούνιο, αποτυπώνονται οι θεσμικές δυσκολίες που υπάρχουν σε σχέση με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και περιλαμβάνεται και η αιρεσιμότητα που πρέπει να πληρωθεί εκ μέρους της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προκειμένου να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ε, θυμίσω για λόγους ιστορικούς ότι ε, το 2003 ακόμη εκκρεμούσε το ζήτημα της ένταξης της Κροατίας που τώρα πλέον είναι το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους επόμενους μήνες γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες που έχουμε συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι περιορισμένες λόγω των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά έχουμε την δυνατότητα να αναλάβουμε πολιτικές πρωτοβουλίες εν ώψη της μεγάλης πολιτικής συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και σίγουρα ένα από τα κεφάλαια της μεγάλης αυτής συζήτησης εν ώψη και των ευρωπαϊκών εκλογών είναι το κεφάλαιο της διεύρυνσης. Επιθυμία μας είναι να προσεγγίσουμε τη διεύρυνση δυναμικά και όπου είναι εφικτό να προωθήσουμε την ενταξιακή διαδικασία επιμέρους χωρών με έναν τρόπο ο οποίος είναι βέβαια προσανατολισμένο σε πρακτικά αποτελέσματα και όχι απλά σε μια ρητορική περιδιεύνησης. Το κρίσιμο είναι η προσήλωση και η δέσμευση των υποψηφίων χωρών στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτήν καθεαυτήν την διβρυσιακή διαδικασία, γιατί αυτό είναι τελικά το κριτήριο. Κάθε χώρα κρίνεται με βάση τις δικές της προσπάθειες και με βάση τον βαθμό προσέγγισης των κριτηρίων που ισχύουν για όλα τα υποψήφια μέλη. Επιτρέψτε μου μια ειδική αναφορά σε σχέση με την Τουρκία εν και τη αυριανή επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού στι Βρυξέλλες και τη συνάντησή του με του επικεφαλεί των θεσμικών οργάνων τη Ένωση. Χαιρετίζουμε το πρόσφατο άνοιγμα του κεφαλαίου 22 που αφορά στην περιφερειακή πολιτική. Είναι όπως ξέρετε καλύτερα από μένα το 14ο κεφάλαιο που ανοίγει από το 2005 όταν ξεκίνησαν οι ενταξικές διαπραγματεύσεις και το πρώτο μετά από τρία και πλέον χρόνια στασιμότητας. Βεβαίως είναι προφανές ότι όλα κρίνονται στα βασικά και θεμελιώδη κριτήρια της ένταξης άρα σίγουρα για την Τουρκία πολύ μεγάλη σημασία έχει η τρέχουσα πολιτική και θεσμική κρίση να εξελιχθεί με έναν τρόπο συμβατό με τις ευρωπαϊκές αξίες. Και προφανώς πρέπει να αναφέρω ότι η εξελίξεις στην Κύπρο, η στάση της Τουρκίας σε σχέση με την επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι, σύμφωνα με τα υφιστάμενα κριτήρια της Κοπεχάγης, ένα σημείο στο οποίο θα κριθεί η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι δυστυχώς η Τουρκία αρνείται όχι απλώς να αναγνωρίσει αλλά ακόμη και να δεχθεί την ύπραξη ενός από τα 28 κράτη-μέλη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά υφίστανται πολλά και σημαντικά κεφάλαια η πρόοδος επί των οποίων εξαρτάται από ζητήματα τα οποία δεν είναι τόσο κρίσιμα όσο αυτά που προανέφερα. Είναι κεφάλαια που αφορούν πεδία πολιτικής στα οποία μπορούν να γίνουν βήματα έτσι ώστε να υπάρχει πάντα ένας ρυθμός, ένα momentum σε σχέση με την ενταξιακή πορεία, με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Για μας η ευρωπαϊκή Τουρκία, η θεσμικά και πολιτικά σταθερή Τουρκία είναι πάντα ένα μεγάλο ζητούμενο και μια βασική προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Τέλος, για λόγους πληρότητας να σημειώσω ότι ως προς την Ισλανδία προφανώ λάβαμε υπόψη μα την απόφαση τη ίδια τη Ισλανδική κυβέρνηση για αναστολή των διαπραγματεύσεων. Εξακολουθούμε φυσικά να συνεργαζόμαστε με την Ισλανδία σε μία σειρά θεμάτων στο πλαίσιο τη συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στο σύστημα Σέγγεν. Θα μου επιτρέψετε να σταματήσω στο σημείο αυτό, αφήνοντας αρκετά επιμέρους ζητήματα για την συζήτηση, στην οποία θα ήθελα αν και εσείς συμφωνείτε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο από τον μονόλογο των εισαγωγικών παρατηρήσεων. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχετε κάνει ένα σφάλμα, έχετε δώσει έναυσμα σε πολλούς ομιλητές να ζητήσουν το λόγο. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Έχουμε 18 μιλητές οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο. Για να μπορέσουμε να έχουμε και απαντήσεις, σας παρακαλώ να είσαστε όλοι σύντομοι και να αυτοπεριοριστείτε χρονικά. Θέλω να τονίσω ότι η απόφαση του Συμβουλίου για την Ουκρανία δείχνει ότι υπάρχει μια γενική δυσκολία για την πολιτική μας γειτονίας. Γιατί δειχθήκαμε όχι ικανοί να θεμελιώσουμε μια κοινή πολιτική έναντι της ε, Ρωσίας. Δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά είναι θέμα της αδυναμίας πολλών κρατών μελών να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική πλήρως και να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε μια κοινή θέση στα θέματα αυτά. Αυτό δεν αποτελεί μια πολιτική αντιρωσική, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να ληφθεί στα σοβαρά όσο δεν έχει μια ενιαία πολιτική κατά έναντι της Μόσχας. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί πέραν των επιμέρους ερωτήσεων. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι σαφές και όταν ήμασταν στην Αθήνα και είναι η επίσκεψή μας, ότι τα θέματα της Μεσογείου και ιδίω της Ανατολικής Μεσογείου είναι πολλά θέματα τα οποία δεν έχουμε λάβει υπόψη επαρκώς με σοβαρότητα. Τα θέματα του δικαίου της θάλασσας συνδέονται με υποβόσκουσες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα θέματα της εξόρυξης φυσικού αερίου, οι διαφορές μεταξύ Κύπρου, Λιβάνου, Ισραήλ, Τουρκίας, όλα αυτά διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αν δεν μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στα θέματα αυτά, όχι μόνο θα χάσουμε χρήματα, θα χάσουμε και την ενεργειακή ασφάλεια την οποία επιζητούμε, αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε και περαιτέρω εντάσεις. Ξέρετε τώρα ότι στο Λίβανο η Χεσμολά θέλει να αλλάξει την οριοθέτηση της, ε, των θαλασσίων ζωνών, κάτι το οποίο οδηγεί σε συγκεκριμένες ανησυχίες για θέματα ασφάλειας. Και επομένως αυτά είναι θέματα για τα οποία ενδεχομένω εμείς ως Επιτροπή θα μπορούσαμε να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη αντιμετώπισης της και να κάνουμε και μια πρόταση κατά τη διάρκεια της ε, ελληνικής προεδρίας που ενδεχομένως θα θέλει να τα υποστήριξει όλα αυτά τα θέματα. Ο κ. Σαλαφράκα έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να σας καλωσορίσω εδώ και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο κατά τη διάρκεια της εξάμενης προεδρίας σας. Ελπίζω ότι καλές προοπτικές της ομιλίας του Πρωθυπουργού σας να γίνουν πραγματικότητα. Αφγανιστάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει βέβαια και καταδικάζει την επίθεση με αποτέλεσμα θύματα δύο μελών μεταξύ άλλων της Ευρωπαϊκής Αποστολής. Εσείς τονίζετε τα θέματα της ασφάλειας και υπογραμμίζετε την αναγκαιότητα να ολοκληρωθεί η συμφωνία εκείνη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Αφγανιστάν προκειμένου να επιβεβαιωθεί η Συμφωνία Ανάπτυξης και Συνεργασίας. Πιστεύετε ότι κατά διάρκεια της Προεδρίας σας θα γίνει αυτό. Δεύτερον, Σύρια. Η Γενέβη 2 αρχίζει την Τετάρτη με συμμετοχή του Ιράν. Τι προπτικές βλέπετε εσείς σε σχέση με τις πτυχές που ανέφερε το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του, δηλαδή προσωρινή κατάπαυση του πυρός, να αντιμετωπιστούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, να απελευθερωθούν κρατούμενοι κλπ. Θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι δικές σας εντυπώσεις γι' αυτό. Και τέλος, το τελευταίο σημείο, αναφερθήκατε στην Ουκρανία και είπατε ότι η έγκριση του νόμου αυτού από την Ράντα κατέδειξε ότι το χάσμα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα αυτή μεγαλώνει. Την επόμενη εβδομάδα μία αντιπροσωπεία ντόκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα επισκεφθεί την Ουκρανία. Θέλω να ξέρω τι προτάσεις έχετε να κάνετε, δηλαδή τι θα θέλατε εκ μέρους της Ευρώπης να μεταφέρουμε εκεί. Και θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας η επόμενη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης να λάβει χώρα στην Ελλάδα. Ε, ε, κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Είναι κάτι που όλοι περιμένουμε, την, ε, τον ηγετικό ρόλο αυτό της Ελλάδας, όμως επειδή η γειτονία μας και ο κόσμος μας ε, σε συνδυασμό με τη δική μας εσωτερική κράση, κρίση καταραίουν, περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Ήθελα να ρωτήσω τα εξή. Αναφέρατε την ανησυχία σας και τον ενδιαφέρον σας για μια ενιαία θαλάσσια πολιτική. Ποια είναι η δική σας θεώρηση γι' αυτό και πώς θα μπορούσε να συνδυαστεί με την απόφαση του ΟΗΕ για την καταστροφή ε, των χημικών όπλων από τη Συρία σε μια περιοχή που είναι στα ανατολικά της Κρήτης και της Μάλτας. Ε, αυτό, αυτή η διαδικασία πώς ε, επηρεάζει τη δική σας θεώρηση για την ενιαία θαλασσία πολιτική. Επίσης στη Συρία. Εγώ έχω δει τον εικονικό αυτό πόλεμο μεταξύ Ιράν και Σαδικής Αραβίας εκτός από από τα εσωτερικά τους προβλήματα να εκτελήσετε και αλλού. Και να εμπλέκετε και το Ιράκ, δηλαδή πέραν των εσωτερικών προβλημάτων, να συμπαρασύρετε το Ιράκ. Τι θα κάνετε εσείς για αυτή τη διαδικασία επιτάχυνσης της διάλυσης του Ιράκ από ό,τι φαίνεται, για την Τουρκία. Σημειώνω όσα είπατε. Όμως, τι μήνυμα αποστελέτε εσείς προς τον Πρωθυπουργό Ερντοάν, διότι πράγματι τα μέτρα για τον δικαστικό κλάδο και ο διαχωρισμός, η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι που θα πλησιάσει ή θα απομακρύνει την Τουρκία από τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Για την Κύπρο επίσης πιστεύετε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από όσα γίνονται στην Τουρκία. Και τι ε, θα πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει από την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Θα περιμένουμε πρώτα να γίνει γενοκτονία και μετά να υπάρξει παρέμβαση. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, ανοίξατε πολλά θέματα και νομίζω το Συμβούλιο ε, είχε υπερβολικά πολλά σημεία στην ημερήσια μεταξύ του. Νομίζω καλύτερα θα ήταν να τα ήταν λιγότερα γιατί πραγματικά έτσι διαχειρίστηκε κάπως η προσοχή του και ίσως δεν ήταν τόσο μεγάλη και αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο τρόπος που θα προβληθεί αυτό εξωτερικά. Θέλω να επικεντρωθώ σε ένα ζήτημα εγώ στην Ευρώπη είδαμε νέα φαινόμενα φοβίας προς την Τρόικα, η οποία έχει ταυτιστεί με ότι είναι αρνητικό, κακό ή απαράδεκτο για τις διάφορες χώρες, ιδίως αυτές που ζουν δυσκολίες. Η Τρόικα στην Ελλάδα ε, ενίσχυσε τον ευρωσκεπτικισμό, όχι μόνο στη δική σας χώρα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα περιμένουμε και τις ευρωεκλογές, μέσα στη χρονιά. Πώς, ε, Υπουργέ, θα ορίζατε το τι έγινε, τι πήγε στραβά, με δύο λόγια από τη δική σας την ε, εμπειρία, τι πήγε στραβά με την Τρόικα στην Ελλάδα για να μπορούμε να το πούμε κι εμείς ε, στους δικούς μας ψηφοφόρους. Και το άλλο μου ερώτημα είναι για την πρώην Γεγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θεωρώ ότι έχετε τώρα μια ευκαιρία ως Ελλάδα στα χέρια σας, ως ε, ε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να λύσετε το πρόβλημα αυτό, διότι υπάρχουν ε, πολλοί παραλογισμοί στην όλη ατμόσφαιρα, αλλά σίγουρα μπορείτε κάτι να κάνετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ελέγχθη, η Ελλάδα είχε αναλάβει την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενδιαφέροντες καιρούς, όταν γίνονται ε, νέες συμμαχίες στην ε, Μέση Ανατολή που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν και αναδύονται νέες, νέες αντιπαραθέσεις μεταξύ χάρη Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Επίσης, η Προεδρία σας καλύπτει το χρονικό διάστημα που θα γίνει τελική συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες που <clears throat> έχει αναλάβει η Ελληνική Προεδρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια στρατηγική και εναντί του Ιράν. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσπαθήσει να επεξεργαστεί μια τέτοια στρατηγική τις επόμενες εβδομάδες. Τα θέματα της περιφερειακής ασφάλειας <clears throat> και της αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας και της μείωσης των εντάσεων στην περιοχή είναι απαραίτητη η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επεσκέφθη το Ιράν πριν από τα Χριστούγεννα και είχαμε τεράστια βοήθεια από την ελληνική πρεσβεία και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Δεύτερον για το θέμα της Ουκρανίας. Η απόφαση του Συμβουλίου λέει ότι είμαστε ανήσυχοι για την κατάσταση στην Ουκρανία. Δεν είναι μονάχα θέμα ανησυχία όμω, είναι πολύ περισσότερο. Η ομάδα των Πρασίνων τουλάχιστον είναι κάτι περισσότερο από ανησυχία. Χρειαζόμαστε πιο έντονου δεσμού με τι χώρε τη εταιρική της ανατολικής εταιρικής σχέσης και με τις πολύπλοκες κοινωνίες τους. Χρειαζόμαστε μια πιο έντονη προσέγγιση προς το λαό της Ουκρανίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήλθατε και τις πιο θερμές ευχές μου για την ε, ελληνική προεδρία από την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Πάρα πολύ αναφέρθηκαν στο θέμα της Ουκρανίας. Εγώ έχω σοκαριστεί από τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε αυτό το πακέτο νόμων που ουσιαστικά ποινικοποιεί την ε, δυσφήμιση, πιέζει τις ε, ελευθερίες έκφρασης και ποινικοποιεί δράσεις των ΜΚΟ. Αν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια καταστολή των ε, ειρηνικών διαδηλώσεων, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κυρώσεις όπως και στη Λευκορωσία κατά της κυβέρνησης αν συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αναφέρθηκε και το θέμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Εγώ χαίρομαι για την αποστολή της ΚΕΠΑ εκεί και επίσης χαίρομαι για την διάσκεψη της Γενέβης 2 για τη Συρία και ελπίζω ότι η Ρωσία θα μπορέσει να ασκήσει κάποια πίεση στην κυβέρνηση του Ασάντ αλλά επίσης και να υπάρξει και πίεση στις χώρες του πεσκού κόλπου για την Αλκάιντα και την ISIS που είναι αποκτούν όλο περισσότερο έδαφος μεταξύ των ε, ανταρτών στη Συρία. Αναφερθήκατε στην ε, Αίγυπτο που υπήρξε 98% υποστήριξη στο νέο Αιγυπτιακό ε, Σύνταγμα. Συζητήθηκε αυτό το θέμα και τι υποστήριξη μπορεί να δώσει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταθεροποιηθεί περισσότερο η Αίγυπτο τόσο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση τη οικονομική ευμάρεια αλλά επίση και για να μπορέσει να προαγάγει περισσότερο τη δημοκρατία, την προστασία των μειονοτήτων, ιδίω των κοπτών. Και ένα άλλο θέμα όπου μπορώ να αναφερθώ σε εσά και ως ε, αντιπρόεδρο τη ελληνική κυβέρνηση. Ξέρω ότι υπάρχει ο μεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος έχει επαφές και με εσά και όχι μόνο με τις δύο κοινότητες. Έχετε κάποιες ελπίδες για μια τομή και μια λύση του προβλήματος κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Οι αποφάσει τη Συνόδου Κορυφή για την άμυνα το Δεκέμβρη του 2013 σηματοδοτούν έξαρση τη επιθετικότητα και τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών εκτός και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημερινή απαράδεκτη απόφαση για την νέα εμπεριαλιστική επέμβαση της Ένωσης στην κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι ακόμα μία απόδειξη. Την καταδικάζουμε αποφασιστικά. Επιδίωξη γενικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική ως παγκόσμιος χωροφύλακας σε συμπλήρωση του ΝΑΤΟ προς όφελος των μονοπωλίων. Εν μέσω τη βαθιά καπιταλιστική κρίση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο ο ανταγωνισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τι άλλε υπεριαλιστικέ δυνάμει για ζώνε επιρροή, έλεγχο τη ενέργεια των σπάνιων γέων και άλλων πρώτων υλών, των οδών μεταφορά για έλεγχο των θαλασσών, του κυβερνοχώρου και του διαστήματο. Στόχο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να επεμβαίνει πιο αποτελεσματικά, πιο γρήγορα, πιο φωνικά, χιλιάδε χιλιόμετρα μακριά από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Γι' αυτό η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, η πιο άμεση αξιοποίηση μάχημων μονάδων, ο έλεγχο των θαλασσών. Θα ήθελα με την ευκαιρία να καταδικάσω επίση την απαράδεκτη απόφαση του Δεκεμβρίου σχετικά με την πολεμική βιομηχανία, που οδήγησαν εκτό των άλλων στη διάλυση των ελληνικών αμυντικών συστημάτων, των ναυπηγείων και τη ΕΛΒΟ, με χιλιάδε απολυμμένου προ όφελο των μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων και των υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Αν συμφωνείτε θα προσπαθήσω να σας περιορίσω σε ένα λεπτό. Οι συντονιστές βέβαια είχαν λίγο περισσότερο χρόνο. Η Μαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχηθώ μια καλή προεδρία στον Πρόεδρο και φίλο κύριο Βενιζέλο. Ε, μας ε, είπε όσα συζητήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής εκεί που ήθελα εγώ να επιμείνω λίγο περισσότερο είναι στις σχέσεις με τη Ρωσία. Δηλαδή πώς προγραμματίζεται αυτή η συνάντηση που θα γίνει στις 28 του μηνός και ποιες ελπίδες έχουμε να βρεθεί κάποιος μέσος δρόμος με τη Ρωσία όπως είπατε και εσείς και να φανεί αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ουκρανία και στη Γεωργία και γενικότερα στην πολιτική γειτονίας που φαίνεται να μην καταλήγει εκεί που θέλαμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κύριο Βαγγέλη Βελιζέλο και να ευχηθώ το καλύτερο για την ελληνική Προεδρία. Ε, ήταν πάρα πολύ αναλυτικός ε, και στις προτεραιότητες και στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Θέλω να κάνω μόνο δύο πολύ συγκεκριμένα. Το ένα είναι για το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό είναι σε πολύ κρίσιμη στιγμή. Λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε όμως ε, σχέδιο για οικοδόμηση 1.800 νέων κατοικιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Πώς σκέφτεται το Συμβούλιο να αντιδράσει σε αυτό. Και δεύτερη και τελευταία ερώτηση. Κύριε Βενιζέλο, είσαστε αισιόδοξο για τη λύση του Κυπριακού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για την Ουκρανία ανέφεραν ήδη πολλοί συνάδελφοι την άποψή της για την κατάσταση τις τελευταίες μέρες και θέτω φυσικά και εγώ το ερώτημά μου αν εντυπωσιάζεται ο κύριος Γιαννουκόβιτς όταν εμείς αποφασίζουμε απλώς ότι θα παρακολουθήσουμε τις ε, εξελίξεις και θα προσαρμόσουμε τις στάσεις μας. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να έχει κάποια επίδραση εκεί είναι αν όλα τα κράτη-μέλη ζητήσουμε με στοχοθετημένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει και την μετακίνηση χρημάτων από άτομα και επιχειρήσεις. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ε, κατάλληλες ε, ενέργειες ώστε να πληροφορούνται τα κράτη-μέλη για τις έρευνες οι οποίες γίνονται γιατί υπάρχουν και μεγάλα ποσά τα οποία έχουν βρεθεί εκτός της Ουκρανίας και αυτό είχε να κάνει με την ε, τήρηση των ε, διεθνών υποχρεώσεων της χώρας αυτής, οι οποίες έχουν παραβιαστεί. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Υπουργέ, σα καλωσορίζω με τη σειρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εύχομαι ολόψυχα μια επιτυχή προεδρία στην Ελλάδα. Ε, μια Προεδρία που απολογισμό τη να είναι ισχυροποίηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνέ γίγνεσθε. Και μια Προεδρία που θα παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και μιλώντα για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ε, κύριε Υπουργέ, με οδηγεί στην ερώτηση και το ζήτημα που θέλω να σα θέσω. Ε, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2003, αναθεωρήθηκε το 2008. Έκτοτε το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας έχει δραματικά αλλάξει. Όμως δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες απειλές και στις νέες προκλήσεις το δόγμα, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας. Βλέπω ότι στο εξάμεινο που θα σκίσει η χώρα σας την Προεδρία, που θα σκίσει η Ελλάδα την Προεδρία, προβλέπεται να υιοθετηθεί ή εν πάση περιπτώσει να γίνει μια ουσιαστική πρόοδος στο να υπάρξει ένα, μια ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας που θα είναι σαφώς μια προστιθέμενη αξία και μια σοβαρή βελτίωση και μια προστίκη σε ένα κενό που πράγματι υπάρχει. Διότι η θαλάσσια πτυχή της ασφάλειας δεν είχε καλυφθεί στις δύο προηγούμενες προσπάθειες να παρουσιαστεί ένα δόγμα ευρωπαϊκής ασφάλειας πέραν ίσως της πειρατείας. Πώς το βλέπετε αυτό και αν πιστεύετε ότι στην Προεδρία θα υπάρξει χρόνος ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Λίζεκ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα κι εγώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Μπροκ και η κυρία Γιαννάκου, ότι δηλαδή το Αφγανιστάν, η Συρία είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και οι Συριανοί σημαντικά θέματα γιατί έχουν άμεση επίπτωση στην παγκόσμια ειρήνη. Πιστεύω όμως ότι είναι απογοητευτικό ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων δαπανά τόσο χρόνο στα, σε άλλα θέματα και δεν λαμβάνει υπόψη αυτά που γίνονται πολύ κοντά στα σύνορά μας τα ευρωπαϊκά. Θα πρέπει να βάλουμε τα του οίκου μας σε τάξη προτού αντιμετωπίσουμε παγκόσμια θέματα. Και αναφέρομαι προφανώς το θέμα της ανατολικής εταιρική σχέσης, τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα και τη ρωσική πολιτική εναντί κρατών. Δεν θεωρείτε κύριε Υπουργέ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών αποκλειστικά αφιερωμένη στο να αντιμετωπιστεί το θέμα της ε, ανατολικής γειτονία τη Ευρωπαϊκή ε, Πολιτική και την σχέση αυτών των χωρών με τη Ρωσία. Ο κύριος Μπουτικόφερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλήρης θεμάτων. Έχετε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αναφέρατε. Αναρωτιέμαι όμως αν μπορούμε να έχουμε σαφήνεια σε σχέση με τις προτεραιότητές μας και να δούμε καλύτερα ποιες είναι οι κεντρικές γραμμές της πολιτικής μας. Στην Frankfurter Allgemeine υπήρχε μία εκτίμηση των διατλαντικών σχέσεων και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αποξενωνόμαστε, ότι υπάρχει μια αυξανόμενη κρίση σε διατλαντικό επίπεδο. Αν έρθει ο πρόεδρος Ομπάμα το Μάρτιο, θα μπορέσετε να θέσετε αυτό το ερώτημα. Είναι στόχος της Προεδρίας σας να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις εντάσεις οι οποίες αναδύονται στην από Ανατολή και αν η Ευρώπη θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της μονάχα στην άμεση γειτονιά της και τα ευρύτερα παγκόσμια θέματα να τα αφήσει σε άλλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θίξατε πολλά θέματα. Θα περιοριστώ μόνο σε ερωτήσεις όπως και οι άλλοι συνάδελφοι. Όχι γιατί τα αφήσατε εσείς, μάλλον έχω ασάφειες σε αυτά που είπατε, αλλά μάλλον κάποιες πλευρές που, που με ενδιαφέρουν ίσως δεν προλάβατε να τις δείξετε. Συρία, ερώτηση πρώτη. Στις διαπραγματεύσεις θα αντιπροσωπευθούν όλοι οι πολιτικοί, κοινωνικοί, εθνικοί φορείς στη Συρία. Παραδείγματο χάρη οι Κούρδοι τη Συρία που είναι το 15% έχουν συμμετοχή εκεί. Και δεύτερη ερώτηση για το θέμα τη Συρία. Αληθεύει το γεγονό ότι η ταφή των χημικών αποβλήτων, κύριε Πρόεδρε, θα γίνει ανοιχτά τη Κρήτη. Και δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με τι προτεραιότητε τη Ελληνική Προεδρία και ειδικά με το μεταναστευτικό. Γνωρίζετε ότι επί τη προηγούμενη ελληνική προεδρίας υπεγράφει το Δουβλίνο 2. Τώρα έχουμε το Δουβλίνο 3. Θα εφαρμοστεί από το Φεβρουάριο του, του του έτους. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση κύριε Πρόεδρε. Έχει συγκατατεθεί δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση στο Δουβλίνο 3 που από όσο ξέρουμε δεν έχει ικανοποιήσει, δεν έχει άρει τα προβλήματα που δημιούργησε το Δουβλίνο 2. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα όλες μου τις ευχές για την Προεδρία σας. Αναφερθήκατε λίγο στην Κύπρο. Κατά τη γνώμη μου, τώρα υπάρχει ένα έβρος ευκαιριών. Η δικιά σας η Προεδρία θα μπορούσε να είναι ιστορική σημασίας αν καταφέρνατε να λύσετε το θέμα και να υπάρξει επανενοποίηση της νήσου. Για την Τουρκία. Το μόνο που είπατε είναι το νόμο Κουλεκή. Αναφερθήκατε επίσης στην διάκριση των εξουσιών. Θέλετε να συμβουλέψετε επίσης την Τουρκία να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα ώστε να μην πάει πιο πίσω η κατάσταση, να μην οπισθοχωρήσει. Για την Ουκρανία επίσης μας είπατε δύο λόγια. Βρίσκεται όμως δίπλα μας. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη δράση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να συμφωνήσω με την προλαλή σας. Ένα θέμα θέλω να αναφέρω και εγώ, την Ουκρανία. Το Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ για τις εξελίξεις εκεί, πως απομακρύνεται από τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία η χώρα. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι έχουμε δουλέψει τόσο πολύ για τη συμφωνία αυτή σύνδεσης, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει ο κόσμος να δει ότι θετικά προχωράει και εξελίσσεται η υπόθεση αυτή. Άρα χρειάζονται συγκεκριμένα βήματα. Κάτι παραπάνω συγκεκριμένο να μπορούμε να πούμε στον κόσμο πέρα από το ότι ανησυχούμε. Οπότε ρωτάω, τι συνέχεια θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο με τον οποίο το καθεστώς ε, Γιαννουκόβιτς προχωράει που τελικά οδηγεί τη χώρα σε ένα δικτατορικό ουσιαστικά καθεστώς μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Υπουργέ, ε, πρέπει να πετύχει η Προεδρία και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Νομίζω ε, καλωσορίζουμε που ήρθατε εδώ πέρα. Ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ασκήσει κριτική για τον τρόπο που γίνονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών για τις εμπορικές σχέσεις. Και έχει ζητήσει να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχει και παρουσία της κοινωνίας των πολιτών και του Κοινοβουλίου. Τι θα κάνει γι' αυτό το Συμβούλιο. Δεύτερο, είναι σχετικό. Ο Σνόουντεν μας άνοιξε τα μάτια για τις μαζικές παρακολουθήσεις ε, όμως τιμωρείται. Και αυτό είναι ένα κακό μήνυμα προς όσους πραγματικά αποκαλύπτουν την υπέρβαση νομιμότητας από τους κρατικούς φορείς. Είναι έτοιμο το Συμβούλιο να κινήσει μια συζήτηση για άσυλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Νόντεν. Το τρίτο, κλιματική αλλαγή. Το Μάρτιο του 2014 πρέπει το Συμβούλιο Υπουργών να αποφασίσει στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα 2030 αλλά και για την μετά Κιώτο εποχή. Είναι προετοιμασμένη η ελληνική προεδρία ε, για αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητά συγκεκριμένου στόχου. Και για τα χημικά όπλα τη Συρία συμμετέχει το Συμβούλιο, έχει πληροφόρηση το Συμβούλιο γιατί το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί οι πολίτε ανησυχούν αλλά δεν έχουμε πληροφόρηση, ούτε το Κοινοβούλιο. The Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τις ευχές που διατυπώσατε προς την ελληνική Προεδρία προκειμένου να πετύχει στις προτεραιότητές της και στους θεσμικούς στόχους της. Επίσης σας ευχαριστώ για τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίο μου θέσατε πολλές ερωτήσεις αλλά όλες είναι αυτονόητες και προφανούς αξίας μετά τα όσα είχα και εγώ τη τιμή να σας πω ενημερώνοντάς σας για τα όσα διημήθησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Ήμουν πράγματι αναλυτικός στην ενημέρωση για τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων γιατί ενεργό εμπροκειμένο εξ ονόματος της μονίμου της υψηλής αντιπροσώπου της κυρίας ε, Άστον και έτσι είχα την υποχρέωση να διαβάσω ένα κείμενο στα αγγλικά προκειμένου να μην κάνω καμιά δική μου παρερμηνία ή παρέκβαση. Ε, ήμουν πιο συνοπτικός στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας γιατί γνωρίζω πολύ καλά το περιθώριο, το στενό περιθώριο μέσα στο οποίο κινείται η εκάστοτε περιοδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πέμπτη ελληνική προεδρία μετά την ένταξη της Ελλάδας στις τότε ευρωπαϊκές κοινότητες το 1981. Προσωπικά είχα την τύχη να μετάσχω ως υπουργό σε άλλες δύο προεδρίες, αυτή είναι η τρίτη προεδρία. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η προεδρία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, ούτε μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τις μόνιμες προεδρίες και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Eurogroup που είναι ένας σχηματισμός ενισχυμένης συνεργασίας, είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη της τις ευαισθησίε όλων των κρατών μελών, έναν εσωτερικό συσχετισμό δυνάμεων που δεν είναι μόνο διαθεσμικός, αλλά είναι είτε το θέλουμε είτε όχι και διακυβερνητικό, ιδίω στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα θέματα κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας. Ε, θα επιχειρήσω λοιπόν να απαντήσω εξηγώντα πού σας λέω την άποψη της ελληνικής κυβέρνησης και της ελληνικής προεδρίας και πού τη θέση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Το ζήτημα της Ουκρανίας πράγματι μας απασχολεί σε όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες. Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων είναι κυλιόμενη. Κάθε μήνα συζητάμε σχεδόν όλα τα θέματα η Ουκρανία, η Συρία, η Αίγυπτος είναι μόνιμα θέματα κάθε συνεδρίασης. Στην Ουκρανία λοιπόν. Πράγματι η πολιτική του διλήμματος ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τη Ρωσία δεν απέδωσε καρπούς. Και δεν απέδωσε καρπούς γιατί το πραγματικό δίλημα που είχε να αντιμετωπίσει η Ουκρανία την περίοδο της Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους κατά τη δική μου άποψη δεν ήταν το δίλημα ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πορεία ή την επιστροφή στη στενή σχέση με τη Ρωσία, αλλά το δίλημα εάν θα βρει τη σωτηρία της εν ώψη της επαπειλούμενης δημοσιονομικής κατάρρευσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή σε κάποιον άλλον που θα σπεύσει να τη βοηθήσει. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα έπρεπε να σημειώσουμε την επομένη του Βίλνιους ήταν το γεγονός ότι η ρωσική κυβέρνηση, ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν, απεφάσισε να αγοράσει ουκρανικά ομόλογα ύψους 15 δισεκατομμυρίων και έτσι να σώσει από μια δημοσιονομική καταστροφή την Ουκρανία με ό,τι αυτό σημαίνει για τους διεθνοπολιτικούς συσχετισμούς στην περιοχή. Υπό την έννοια αυτή η ελληνική προεδρία που διαδέχθηκε τη Λιθουανική βεβαίως και έχει υποχρέωση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Βίλνιους και θα τις εφαρμόσουμε. Βεβαίως και στο επίπεδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα οργανώσουμε μια από τις επόμενες συνόδους μας με βασικό αντικείμενο την ανατολική εταιρική σχέση όπως έχουν ζητήσει πολλά κράτη-μέλη. Βεβαίως και υπό το φως του Βίλνιους και των εξελίξεων στην Ουκρανία επανεξετάζουμε την στρατηγική μας σχέση με τη Ρωσία και προετοιμαζόμαστε για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας στις 28 Ιανουαρίου. Αλλά πρέπει να δούμε με ευθύτητα και ειλικρίνεια εάν μπορούμε να συνεχίσουμε σε μια πολιτική διληματικού χαρακτήρα ή αν πρέπει να κάνουμε μια προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη της μια πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί και η οποία στην πραγματικότητα μας επιβάλλει πριν αξιολογήσουμε την ανατολική εταιρική σχέση να αξιολογήσουμε και να επανατοποθετήσουμε την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Εάν δεν προηγηθεί η αποσαφήνιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής σε σχέση με τη Ρωσία, θα έχουμε αντιφάσεις και ανεπάρκειες σε όλη μας στρατηγική, όχι μόνο σε σχέση με την Ουκρανία, αλλά σε σχέση με όλες τις χώρες που μετέχουν στην Ανατολική γειτονία. Και με τη Γεωργία και με την Αρμενία και με τη Μολδαβία και με το Αζερβαϊτζάν. Άρα αυτό είναι που προέχει. Αυτό το συζητήσαμε σήμερα στο γεύμα εργασία και το είχαμε συζητήσει και τον Δεκέμβριο παρουσία του κυρίου Λαυρόφ σε ένα πολύ ωραίο γεύμα εργασία. Ε, η αλήθεια είναι ότι η στρατηγική μας σε σχέση με τη Ρωσία είναι θύμα μιας πολύ μεγάλης εσωτερικής αντίφασης. Γιατί η κοινή ευρωπαϊκή θέση στο ζήτημα αυτό είναι κατώτερη από το άθροισμα των πολιτικών που ασκούν όλα τα κράτη-μέλη σε διμερές επίπεδο με τη Ρωσία. Η εσωτερική αντίφαση φαίνεται πάρα πολύ καθαρά στο γεγονός ότι εκ των πραγμάτων, de facto, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχεται την προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στα μεγάλα εθνικά θέματα όπου έχουμε σημαντικές κοινέ πρωτοβουλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Αυτό έγινε και στη Συρία και στο Ιράν. Στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει και με την Ουκρανία, Μιλάμε με έναν αφηρημένο τρόπο, αλλά ξεχνούμε να αναφέρουμε ότι η Ουκρανία, όπως και η Ρωσική Ομοσπονδία, είναι εδώ και πολλά χρόνια πλέον μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε μια πολιτική που περικλείει και τους θεσμούς του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Στα θέματα της ενεργειακής πολιτικής των επενδύσεων, των ρωσικών επενδύσεων στην Ευρώπη, της επιχειρηματικής παρουσίας ευρωπαϊκών κρατών στη Ρωσία, όλοι κινούνται σε ένα διμερές επίπεδο. Όλοι θέλουν να διαφυλάξουν παραδοσιακά προνόμια ή να κάνουν μια νέα τοποθέτηση, ένα νέο positioning μπροστά στα νέα δεδομένα, αλλά όχι στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα τα ζητήματα ξεκινούν από εμά. Εμείς πρέπει να ενοποιήσουμε τη στρατηγική μας εμείς πρέπει να αποσαφηνίσουμε το στρατηγικό πλαίσιο Ευρώπης-Ρωσίας για να ξαναδούμε σοβαρά την, Ευρω... την... Ε, την ανατολική εταιρική σχέση. Αλλιώς νομίζω ότι κάνουμε μια επιπόλαιη και αναποτελεσματική προσέγγιση. Θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα. Υφιστάμε τα κάτι μέλη πάρα πολλές πιέσεις στην ενεργειακή μας πολιτική στο όνομα του, δικαίου του ανταγωνισμού και της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε υποστεί πάρα πολλέ πιέσεις σε σχέση με, ε, την, το πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης σημαντικών δημοσίων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική στα θέματα ανταγωνισμού στον τομέα της ενεργειακής αγοράς, αλλά κανείς δεν θέτει το μεγάλο θέμα που είναι να διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τιμές του φυσικού αερίου με την Gazprom με ενιαίο τρόπο. Μα η διαφοροποίηση τη τιμή του φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας είναι για την ελληνική οικονομία εξίσου σημαντική με την διαφοροποίηση των επιτοκίων χορηγήσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε ακριβότερο χρήμα για τις επιχειρήσεις μας και ακριβότερη ενέργεια για τις επιχειρήσεις μας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα να ανορθώσουμε την πραγματική οικονομία. Αυτό δεν είναι αφηρημένη γεωπολιτική. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που συνδέεται με την κατάσταση της οικονομίας σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα νοικοκυριά. Άρα αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, το μεγάλο θέμα σε σχέση με την Ουκρανία και σε σχέση με τη Ρωσία. Και βεβαίως περιμένουμε, δεν είναι δικό μας ζήτημα αυτό, είναι ζήτημα των μονίμων προεδριών, το πώς θα οργανωθεί και τι περιεχόμενο θα έχει η Σύνοδος Κορυφής, Αλλά σίγουρα η Σύνοδος Κορυφής πρέπει και συμβολικά, οργανωτικά να αποτυπώνει την σημασία που αποδίδουμε στη σχέση μα με την ε, Ρωσία. Εξίσου σημαντικό είναι βέβαια να αποτυπώνεται και ο ευρωατλαντικός χώρος και ο ευρωατλαντικός διάλογος. Δηλαδή και η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να έχει πάρα πολύ βαρύνουσα σημασία. Και εκεί φυσικά τα θέματα τα χειρίζεται πρωτίστως η Επιτροπή, αλλά και εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η συζήτηση για το TTIP, η συζήτηση δηλαδή κυρίως για το νέο πλαίσιο συνεργασίας μας ε, στον, στον ευρύτερο χώρο της ε, διεθνούς αγοράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και τις θεσμικές παραμέτρους οι οποίες ούτως ή άλλως ε, απορρέουν από το γεγονός ότι μετέχουμε στον ΠΟΕ, ότι μετέχουμε στον ΝΑΤΟ και ούτω καθεξής. επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στα θέματα τα πιο επίκαιρα της Συρίας. Το μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε στο Συμβούλιο σήμερα ήταν αν η πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα προς το Ιράν να μετάσχει και αυτό στη Γενέβη 2 μεθαύριο δημιουργεί προβλήματα ή μπορεί να προκαλέσει την άρνηση της μετριοπαθούς αντιπολίτευσης να εφαρμόσει την απόφαση που πήρε στην Κωνσταντινούπολη πριν από λίγες μέρες και να μετάσχει στην διάσκεψη. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω πάρα πολύ σύντομα ποια ήταν η παρέμβασή μου στο Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό. Πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος, την αξιοπιστία και την νομιμοποίηση της διαδικασίας αυτής. Δεν πρέπει να δώσουμε καμία εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαφωνεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είναι ο συγκαλών την διάσκεψη, ο οικοδεσπότης και ο θεσμικός εγγυητής της διάσκεψης. Και δεν πρέπει να αφήσουμε την μετριοπαθή Συριακή Αντιπολίτευση να υπαναχωρήσει και να μην έλθει πρέπει να έλθει, οπωσδήποτε. Γιατί χωρίς αυτήν φυσικά δεν υπάρχουν οι συνομιλητές, οι ελάχιστοι δυνατοί συνομιλητές. Εκπροσωπούνται όλες οι πτέρυγες, όλες οι οντότητες, όλοι οι παράγοντες, όλες οι εθνοτικές, θρησκευτικές και πολιτικές ομάδες, όλες οι μαχόμενες ομάδες. Όχι, δεν εκπροσωπούνται. Εκπροσωπείται ένα τμήμα της μετριοπαθούς αντιπολίτευσης, η οποία όμως αναγκάζεται να μετέχει σε έναν πόλεμο μέσα στον πόλεμο στην Συρία. Αλλά αυτή η μετριοπαθή αντιπολίτευση είναι ο πυρήνας από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Άρα πρέπει να διασώσουμε τη διαδικασία, πρέπει να προφυλάξουμε τη σχέση μας, την τριγωνική σχέση Ηνωμένα Έθνη, Ηνωμένε ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαφυλάξουμε και τη σχέση μας με τη Ρωσία χωρίς την οποία και χωρίς την πρωτοβουλία Κέρι Λαυρόφ δεν θα ξεκινούσε η διαδικασία αυτή, να θυμηθούμε τις δεσμεύσει από τη Γενέβη 1 και να προχωρήσουμε στη Γενέβη 2. Σε σχέση με τα χημικά, η καταστροφή των χημικών όπλων δεν απασχόλησε το Συμβούλιο γιατί δεν είναι αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Είναι μια επιχείρηση που εκτελείται από τον αρμόδιο διεθνή οργανισμό, τον OPCW δηλαδή, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κρίσιμος είναι ο ρόλος των κρατών που ασκώντας την εθνική τους κυριαρχία αποδέχθηκαν να μετάσχουν με τον έναν ή άλλον τρόπο στην επιχείρηση αυτή. Άρα από πλευράς ευρωπαϊκών κρατών κρίσιμος είναι σίγουρα ο ρόλος της Δανίας που μετέχει στη μεταφορά. Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρίσιμος είναι ο ρόλος της Ιταλίας η οποία διαθέτει λιμένα στην Καλαβρία ο οποίος είναι εξειδικευμένο στη μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών. Κρίσιμο είναι ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών που διαθέτουν το μεγάλο σκάφος που είναι σκάφος εργαστήριο στο οποίο θα γίνει η υδρόληση. Είναι προφανές ότι εμείς ως χώρα δεν θέλουμε η επιχείρηση αυτή να γίνει στην Μεσόγειο. Διότι η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα. Είναι πολύ πιο λογικό και πολύ πιο ασφαλές αυτό να γίνει στον Ατλαντικό και υπάρχει ετοιμότητα της πορτογαλικής κυβέρνησης να διαθέσει στι Αζόρες λιμάνι για την μεταφόρτωση, ώστε μετά να γίνει η υδρόληση. Βέβαιο όμω είναι, από τη διερεύνηση που κάναμε και από τις συζητήσεις που είχαμε με άλλες κυβερνήσεις, εμπροκειμένου με τη γερμανική πλευρά, πως δεν πρόκειται να γίνει καμία απόρριψη υλικού στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα τη υδρόληση θα μεταφερθεί πάλι χερσαία στην Γερμανία κατά πάσα πιθανότητα όπου θα γίνει η καταστροφή σε εξειδικευμένα εργοστάσια, άρα δεν πρόκειται να απορριφθούν απορρίμματα στην Μεσόγειο. Θα απευθύνουμε σχετική επιστολή στον αρμόδιο διεθνή οργανισμό και η κυρία Μπονίνο και εγώ και η Επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα όπως προκύπτει από τις συνεννοήσεις που είχαμε την αρμόδια Επίτροπο η οποία σκέφτεται να αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία ζήτησε από την κυρία Άστον να ενεργήσει εξ ονόματος του Συμβουλίου πρέπει να έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν κινδυνεύει καθόλου το, μεσογειακό περιβάλλον. Και πρέπει αυτήν την εγγύηση να μας την δώσει ο ΟΗΕ και ο αρμόδιος για τα χημικά όπλα οργανισμός. Ως προς τα θέματα που αφορούν ε, την Αίγυπτο. Ε, τα θέματα της Αιγύπτου τα συζητάμε κάθε φορά και βεβαίως αυτό που είπε το Συμβούλιο είναι ότι το βήμα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Είναι σημαντικό να έχει ένα νέο σύνταγμα η συμμετοχή με τα δυτικά δεδομένα μας φαίνεται μικρή αλλά με τα αιγυπτιακά δεδομένα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη και έχει πολύ μεγάλη σημασία να επιμείνουμε σε αυτήν την έννοια της ε, inclusiveness, σε αυτή την έννοια της ε, συνενετικής και συνερετικής διαδικασίας σε σχέση με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της Αιγύπτου. Αλλά πάντως ε, τα συμπεράσματα και οι δηλώσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε σχέση με την Αίγυπτο διαχρονικά από τον Ιούνιο και μετά αποτυπώνουν αυτή την καμπύλη, δηλαδή στην πραγματικότητα πιέζουν ώστε να εφαρμοστεί ο οδικός χάρτης που έχει εξαγγείλει η μεταβατική Αιγυπτιακή κυβέρνηση για την μετάβαση στην ομαλότητα, γιατί ακόμη προφανώς υπάρχει μια εξαιρετική και έκτακτη κατάσταση. Για τα θέματα που αφορούν το Αφγανιστάν ε, στην πραγματικότητα ναι, το Συμβούλιο αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στην υπογραφή της Συμφωνίας Ασφάλειας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αφγανιστάν. Ξέρετε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις και προβλήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το χειριζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα όμως ότι το κύριο φόρουμ στο οποίο συζητείται το ζήτημα αυτό είναι το ΝΑΤΟ και το σχήμα της ISAF στο οποίο μετέχουν ε, σχεδόν το 1 τρίτο των χωρών του ΟΗΕ. Σε σχέση με τα ζητήματα της, ε, ε, του διαλόγου για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ε, είναι προφανές ότι δεν θα βρεθεί καλύτερη στιγμή. Δεν θα βρεθεί πιο έτοιμη για σημαντικές αποφάσεις κυβέρνηση στην Παλαιστινιακή πλευρά και οι συσχετισμοί στο εσωτερικό της Ισραηλινής κυβέρνησης ούτως ή άλλως πάντα ακολουθούν μια πολύ συγκεκριμένη καμπύλη, μια διακύμανση. Υπάρχει ένα momentum μετά από τις τόσες προσπάθειες της εργόδης που κατέβαλε ο κύριος Κέρι και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί. Ε, υπάρχουν παραβιάσεις αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προφανώς υπάρχουν. Το ζήτημα ε, είναι να ξεκινήσει ο διάλογος ή μάλλον να μην διακοπεί ο διάλογος στην αρχή του και να αρχίσει να αποκτά ένα πολύ πιο συγκεκριμένο και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει συνεχώς και υπογραμμίζει την ετοιμότητά της να βοηθήσει οικονομικά με ένα οικονομικό δέλεαρ εντό εισαγωγικών, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι θα έχει διατηρηθεί ο διάλογος και θα έχει επιτευχθεί μια βασική πολιτική συμφωνία. Αυτό είναι όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ ε, δύσκολο. Σε σχέση με το ζήτημα που ε, είναι οξύτατο τις μέρες αυτές της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας, ε, το Συμβούλιο επεφάσισε να μην ενεργοποιήσει τους μηχανι... τους... τις ευρωπαϊκές ομάδες μάχης, τα battle groups, παρότι αυτό ετέθη από ορισμένα κράτη-μέλη. Συμπτωματικά αυτό ετέθη τώρα που το, η ομάδα μάχης είναι κατά βάση ελληνική. Η Ελλάδα διαθέτει 1.100 από τους 1.500 ε, στρατιώτες που συγκροτούν την ομάδα μάχης. Ε, αλλά η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θεωρεί ορθή επιλογή την χρησιμοποίηση των ομάδων μάχης. Ε, αποφασίσαμε να αναλυφθεί ε, πρωτοβουλία να οργανωθεί επιχείρηση στο πλαίσιο της ε, κοινής, πολιτικής, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, συνεργαζόμαστε ως ελληνική κυβέρνηση με την γαλλική κυβέρνηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της ομάδας που θα πάει, η οποία δεν θα έχει ελληνική συμμετοχή καθόλου, αλλά εφόσον ε, προτιμούν να εκπαιδευτούν στο στρατηγείο της Λάρισας που έχει σχετική τεχνογνωσία, είμαστε διατεθειμένοι να το προσφέρουμε σύμφωνα και με την απόφαση του ε, σημερινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, επαναλαμβάνοντας χωρίς να υπάρχει συμμετοχή Έλληνα στρατιώτη στην αποστολή, γιατί δεν υπάρχει και η σχετική εκπαίδευση, ούτε το ζητάει η Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Σε σχέση ε, με το Λίβανο, το μεγάλο θέμα μας ε, είναι να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Ε, και να αναλυφθεί μια πολύ πιο συγκεκριμένη και φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το έχουμε συζητήσει αυτό με τους ε, συναδέλφους μου στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων και με την κυρία Άστον στην προηγούμενη συνεδρίαση, στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου με έμφαση. Είναι επίσης προφανές ότι το Λίβανο είναι συνεχώς θύμα των περιστάσεων και αυτή τη στιγμή έχει πλημμυρίσει από αλλεπάλληλα κύματα προσφύγων στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες τώρα έχουν προσθεθεί οι πρόσφυγες από τη Συρία. Ε, η κατάσταση στο Λίβανο είναι ούτως ή άλλως έκρηθμη και φυσικά συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έγιναν σε σχέση με το συνεχιζόμενο πρόγραμμα, πρόβλημα στο Ιράκ, με τον κίνδυνο διάλυσης ξανά ε, της θεσμικής του υπόστασης. Ε, αυτή τη στιγμή που συζητούμε πραγματοποιείται όμως το Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιράκ στο οποίο την ελληνική προεδρία εκπροσωπεί ο Υφυπουργό Εξωτερικών λόγω της δικής μου παρουσίας εδώ στην Επιτροπή, θεωρώ ότι υπό τις παρούσες περιστάσεις και με τέτοιες πιέσεις, τέτοια έκρηξη βίας στο Ιράκ, το γεγονός ότι πραγματοποιείται το Συμβούλιο Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντικό ως εθάριση και προς την Ιρακινή κυβέρνηση. Σε σχέση τώρα με την διεύρυνση, ε, και πιο συγκεκριμένα με τα Δυτικά Βαλκάνια. Σε σχέση με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η ελληνική Προεδρία θα εφαρμόσει όσα περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ης Δεκεμβρίου, όσα συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 17 Δεκεμβρίου και εγώ ως Πρόεδρος του Συμβουλίου είμαι έτοιμος τις επόμενες μέρες να επισκεφθώ όλες τις πρωτεύουσες της περιοχής και φυσικά θα επισκεφθώ και τα Σκόπια χωρίς ε, να γίνεται καμία διάκριση ή διαφοροποίηση και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ε, ανάμεσα στην Προεδρία του Συμβουλίου και την κυβέρνηση της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Έχω ήδη συναντηθεί δύο φορές από ό,τι που ανάλαβα τα καθήκοντά μου με τον ομόλογό μου της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη. Έχω συναντηθεί με τον αρχηγό του μεγαλύτερου αλβανικού κόμματος που μετέχει στην κυβέρνηση, τον κύριο Αχμέτη, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ελληνική θέση είναι μετριοπαθής και υπεύθυνη. Έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι σεβόμαστε την διαδικασία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε το ρόλο του κυρίου Νίμιτς, είμαστε σε στενή επαφή μαζί του, αποδεχόμαστε ένα σύνθετο όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό δίπλα στον όρο Μακεδονία, αλλά ένα όνομα για κάθε χρήση. Είναι η περιβόητη έννοια του έργο Ένα όνομα για εσωτερική και εξωτερική χρήση η ένσταση ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύνταγμά μας είναι μια ένσταση ακατανόητη για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αλλάζουμε συνεχώς τα εθνικά συντάγματα για να συμμορφωθούμε είτε στο ευρωπαϊκό δίκαιο είτε στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και γενικώ για να συγκροτήσουμε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό συνταγματικό χώρο. Άλλωστε και η συμφωνία της Οχρίδας η οποία είναι διεθνωτική μεταξύ της σλαβικής και της αλβανικής κοινότητας ήταν μια συμφωνία υβριδική, διεθνής και συνταγματική και εκ του πλαγίου άλλαξε το Σύνταγμα. Το ζήτημα όμως δεν είναι το όνομα. Το πρόβλημα για την ενταξιακή προοπτική της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν είναι το όνομα. Το πρόβλημα είναι η γενική εφαρμογή και ισχύ των κριτηρίων της Κοπεχάγης η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η εσωτερική πολιτική κατάσταση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το γεγονός ότι έχουμε μια επίσημη κρατική ιδεολογία, το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα ανοιχτά ζητήματα με άλλες χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα υποψήφια κράτη. Σε σχέση με την Τουρκία, νομίζω ότι θα έπρεπε να επιφυλαχθούμε να ακούσουμε τι θα συζητήσει ο κύριος Ερντογκάν αύριο με τον πρόεδρο Βαν Ρομπάι, με τον πρόεδρο Μπαρόζο, με τον πρόεδρο Σούλτ. Αλλά βεβαίω υπάρχουν τα ευρωπαϊκά κριτήρια τα οποία ισχύουν για κάθε υποψήφια χώρα. Εφόσον η Τουρκία είναι υποψήφια χώρα, πρέπει να πληρεί τα κριτήρια αυτά, να ανταποκρίνεται σε ευαισθησίε και αξίε. Για εμά ω Ελλάδα, σε διμερές επίπεδο, το μεγάλο πρόβλημα είναι να αποφευθεί η λεγόμενη εξαγωγή της εσωτερικής έντασης. Ιστορικά, διαχρονικά, εσωτερικές κρίσεις στην Τουρκία συνδέονται με κρίσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε ανοιχτά κανάλια διπλωματικών επαφών, έχουν αλλάξει εποχές, υπάρχουν σοβαρά ανοιχτά προβλήματα, δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά την εμπειρία της εξαγωγής της εσωτερικής κρίσης. Υπάρχει momentum για το Κυπριακό. Για το Κυπριακό υπάρχει momentum εάν υπάρχει momentum στην Τουρκία. Γιατί ο κρίσιμος παράγοντας για την επίλυση του Κυπριακού είναι η Τουρκία. Δεν το λέω εγώ αυτό. Δεν το λέει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ούτε η ελληνική κυβέρνηση. Το λέει η σταθερή νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που θεωρεί ότι τον έλεγχο στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου το ασκεί η Τουρκία, εναντίον της οποίας ασκούνται οι ατομικές προσφυγές όποιου θίγεται στα θεμελιώδη δικαιώματά του και καταφεύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Άρα η θέση της Τουρκίας είναι τελείως διαφορετική από τη θέση τη δική μας ή οποιοδήποτε άλλου κράτους. Ο διάλογος γίνεται ανάμεσα στις δύο κοινότητες, ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή, αλλά βασίζεται σε ορισμένε αρχές. Ο κύριος Δαβούτογλου και εγώ συμφωνήσαμε η Αθήνα να δεχθεί τον διαπραγματευτή της τουρκοκυπριακής κοινότητας που είναι θεσμική οντότητα του Κυπριακού Συντάγματος του 1960 και η άγκυρα να δεχθεί τον διαπραγματευτή της ελληνοκυπριακής κοινότητας, της κοινότητας, αλλά αυτό θα γίνει αφού συμφωνηθεί το κοινό ανακοινωθέν μεταξύ των δύο ηγετών, των κοινοτήτων και ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Οι προϋποθέσεις αυτονόητες, ο σεβασμός των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και τρεις αρχές που διέπουν κάθε ομοσπονδιακό κράτος. Γιατί πάμε για μια Κύπρο ομοσπονδιακή, διζωνική, δικοινοτική. Ενιαία νομική προσωπικότητα, ενιαία κυριαρχία και ενιαία ηθαγένεια. Και όλα αυτά να γίνουν δεκτά με δημοψήφισμα. Γιατί αν δεν ψηφίσει ο κυπριακός λαός στο δημοψήφισμα δεν υπάρχει λύση. Άρα πρέπει να πάμε σε μια λύση η οποία να μπορεί να γίνει δεκτή με δημοψήφισμα επί τη βάση των αρχών της αυτοδιάθεσης που έχουν γίνει δεκτές ήδη από το 2003 από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ε, και δύο κουβέντες σε σχέση με την ε, Τρόικα και τα ζητήματα τα οποία συνδέονται με την οικονομική κρίση και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Πριν από αυτό να απαντήσω όμως τον κύριο Κουμουτσάκο ο οποίο μου έθεσε ένα πολύ σημαντικό θέμα ευρωπαϊκής Στρατηγική ασφάλειας. Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας μετά την, το 2008 και την αλλαγή του χάρτη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ μας έχει προλάβει το ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ άλλαξε δόγμα στη Σύνοδο Κορυφής τη Λισαβόνας, η οποία συνέπεσε με τη Σύνοδο Κορυφής ΝΑΤΟ ε, Ρωσίας, ε, μετασχηματίστηκε σε έναν οργανισμό ασφάλειας, προσπάθησε να βρει το νέο στόχο, δηλαδή στην πραγματικότητα τη νέα απειλή, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει γίνει με τον ίδιο καθαρό τρόπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό είναι κάτι που ανάγεται στο πώς αντιλαμβανόμαστε ιστορικά την ευρωπαϊκή ασφάλεια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή μετά τους 14 όρους του Προέδρου Wilson και το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση και επί εποχής κοινωνίας των εθνών και επί εποχής Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δύο, δύο, δύο, δύο φράσεις σε σχέση με τα ερωτήματα για την Τρόικα. Γιατί απαντώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τρόικα. Γιατί το ζήτημα της Τρόικας είναι πράγματι ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και κυριαρχίας και ένα ζήτημα θεσμικής ισοτιμίας των κρατών μελών. Η Τρόικα λοιπόν είναι ένα θεσμικό υβρίδιο το οποίο δεν προβλέπεται από τις συνθήκες, τις ιδρυτικές συνθήκες, από το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το κενοφανές στοιχείο. Το κενοφανές στοιχείο είναι ότι μετέχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε μια διαδικασία η οποία είναι ενδοευρωπαϊκή, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αυτό γιατί συνέβη, γιατί δεν υπήρχαν μηχανισμοί διαχείρισης της κρίσης γιατί το εγχείρημα της Ευρωζώνης ήταν κατασκευασμένο για φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως. Άρα λοιπόν οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές ζήτησαν να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να συμβάλλει στη διαχείριση της κρίσης εκφράζοντας την δυσπιστία του στην Επιτροπή. Η Τρόικα είναι έκφραση δυσπιστίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει και μία αλλαγή και διεύρυνση του θεσμικού ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν ασχολείται μόνο με τον καταστατικό της σκοπό, αλλά και με την παρακολούθηση δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών κάποιων κρατών μελών. Δεν ασχολείται μόνο με την νομισματική πολιτική και με τον βασικό σκοπό της που είναι η σταθερότητα των τιμών σύμφωνα με το καταστατικό που τη διέπει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και το θέμα αυτό έχει να κάνει με τον σχεδιασμό των προγραμμάτων προσαρμογής. Όταν στο κατάλληλο φόρουμ το ευρωπαϊκό θα μας δοθεί ευκαιρία να πούμε λεπτομέρειες για το τι έγινε και πώς έγινε, νομίζω ότι θα γίνει πιο εύκολα αντιληπτό αυτό που λέω. Αλλά δεν υπήρχε για μας άλλη καλύτερη λύση. Η λύση που μας επιβλήθηκε δεν ήταν μια καλή λύση, αλλά ήταν η καλύτερη προσφερόμενη λύση. Διότι αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη στην Ευρώπη. Για μας δεν υπάρχει καλύτερο περιβάλλον και καλύτερο εταίρο από την Ευρώπη, από τους Ευρωπαίους εταίρους μας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το δάνειο που μας δόθηκε είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 240 δισεκατομμύρια. Ναι, εάν δεν είχαμε το δάνειο θα είχαμε ασύντακτη χρεοκοπία και κατάρρευση οικονομική, κοινωνική, πολιτική, ίσως και θεσμική. Ναι, έπρεπε να αποφύγουμε την κατάρρευση και να πάμε σε μια συντεταγμένη λύση. Οι όροι που επιβλήθηκαν είναι όροι πάρα πολύ αυστηροί, είναι όροι οι οποίοι απορρέουν από μια ολόκληρη αντίληψη οικονομική, πολιτική, ιδεολογική. αυτό είναι ο εσωτερικό συσχετισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κινούνται όλε οι κυβερνήσει και όλε οι χώρε, γιατί οι συσχετισμοί δεν είναι συσχετισμοί πολιτικοί μεταξύ κυβερνήσεων, είναι συσχετισμοί εθνικών στρατηγικών μεταξύ κρατών μελών και δεν αλλάζουν οι συσχετισμοί αυτοί με την αλλαγή των κυβερνήσεων τόσο εύκολα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο ε, οφείλουμε να το δούμε και το βλέπουμε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι είναι έτσι διαρθρωμένο το πρόγραμμα προσαρμογής ώστε παρά τα λάθη που έχουν γίνει τα κατασκευαστικά από τους σχεδιαστές του του προγράμματος. Παρά τα λάθη τα δικά μας και τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή βέβαια ενός τόσο δύσκολου προγράμματος, υπό κρίσης. Ε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχεις ύφεση 25%. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις ανεργία των νέων 60%. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις απώλεια εισοδημάτων κατά μέσο όρο 35%. Άρα λοιπόν παρά τις δυσκολίες εσωτερικές, παρά τα λάθη των σχεδιαστών του προγράμματος, έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που δεν έχει κοστίσει στον Ευρωπαίο φορολογούμενο ούτε ένα ευρώ. Γιατί το δάνειο εξυπηρετείται, οι εγγυήσει που έχουν χορηγηθεί δεν θα καταπέσουν και μόνο μία περίπτωση υπάρχει να χρειαστεί να πληρώσουν Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Να αποτύχει το πρόγραμμα και να βρεθεί η Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να σεβαστούν τις θυσίες του ελληνικού λαού και να πάψουν να ανακυκλώνουν μια άδικη συζήτηση για το αν η Ελλάδα μπορεί ή δεν μπορεί. Λοιπόν η Ελλάδα μπορεί, το χρέος μας έχει αναδιαρθρωθεί και όσοι μετέχετε σε επιτροπές που έχουν σχετική αρμοδιότητα θα παρακαλούσα να υποβάλλετε τις σχετικές ερωτήσεις στον επικεφαλής του ESM, τον κύριο Ρέγκλιν, για να εξηγήσει αυτός και όχι εγώ πόσο βιώσιμο είναι το ελληνικό χρέος σε όρους καθαράς παρούσας αξίας σε όρους net present value. Γιατί εκεί φαίνεται πόσο μεγάλη ήταν η αναδιάρθρωση και πόσο πιο βιώσιμο είναι το ελληνικό χρέος σε σχέση με το χρέος άλλων κρατών μελών. Πάρα πολύ συνοπτικά αυτή είναι η απάντησή μου, την οποία θα χαιρόμουν σε ένα άλλο φόρουμ ασχολούμενο με τα θέματα οικονομικής πολιτικής να τη δώσω πιο αναλυτικά, όχι ως Υπουργός Εξωτερικών, αλλά ως πρώην Υπουργός Οικονομικών και ως Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δώσατε και για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δει όλοι ότι η Ελλάδα έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να βγει από την κρίση και υπάρχουν σημαντικές πρόοδοι Ελπίζω ότι μέχρι το, τις αρχές του 2015 η κυβέρνηση θα φέρει σε πέρα στη, την πολιτική της για να μπορέσουν να υπάρξουν απτά αποτελέσματα υπέρ του ελληνικού λαού. Σας εύχομαι λοιπόν και σε εσά και στα διακόμματα που βρίσκονται στην κυβέρνηση κάθε επιτυχία. Είναι σημαντικό όχι μόνο για εσάς αλλά και για μας. σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις σας. για την Ουκρανία. Εγώ βρίσκω σημαντικό αυτό το οποίο αποφάσισε το Συμβούλιο που κρατάει ανοιχτή την πόρτα. Δεν ξέρουμε τώρα αν η Ουκρανία κινδυνεύει να πέσει σε μια ρωσική παγίδα. Χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να εκτιμήσουμε την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό κάθε δύο-τρεις μήνες θα πρέπει να έχουμε μια επανεξέταση. Και το ίδιο ισχύει και με τις ενεργειακές τιμές. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα διαμορφωθούν αυτές οι τιμές από το, τα πρώτα χρήματα που πήρε η Ρωσία τα χρησιμοποίησε για την αποπληρωμή παλαιότερων χρέων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε μεγάλη σημασία. θεωρητικά προσπαθεί η Ρωσία να σώσει την Ουκρανία από την κρίση, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε αν οι ενέργειές της έχουν σαν στόχο να την βυθίσουν ακόμα περισσότερο στην κρίση. Αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ελπίζω θα μπορέσουμε να ξανασυναντηθούμε και στο μέλλον. Frage, eine kurze, ja. kurze Dinge vor der Abstimmung. Das Kannst du ihm sagen vielleicht? Ja. Ne? Herren, Ich möchte den Tagesordnungspunkt 10 aufrufen. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης για τον κύριο Τάνοκ. Του προτείνω να λάβει το λόγο διαβραχαίως αύριο πριν από την ψηφοφορία να μας εκφράσει τη θέση του για τις ε, τροπολογίες ε, συμβιβασμού. Νομίζω ότι είναι καλύτερα γιατί πάρα πολλοί σήμερα έτσι άλλως δεν θα είναι παρόντες να τον ακούσουν. Στην αρχή πριν από την ψηφοφορία. Ναι, πράγματι θα λάβω το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να λάβω το λόγο, λέει ο κύριος Στάνο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας, λέει ο πρόεδρος. Και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το επόμενο σημείο. David O'Sullivan ο κύριος Ντέβιτο Σάλιβαν ε, θα λάβει το λόγο και αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης είναι και κλεισμένο το θυρών. Τα ελβετικά τυριά έχουν τρύπες. Η Επιτροπή μας όμως δεν έχει τρύπες.